Okay, let's... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρία της Επιτροπής ε, ασφάλειας και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι προτεραιότητα για τη διερμηνία έχουν μόνο οι γλώσσες των πλήρων μελών. Άρα ε, με τα λύπη μου θα σας πω ότι δανέζικα, λιθουανικά, σουηδικά, λετονικά, σλοβακικά, βουλγάρικα, ε, τσεχικά και ουγγρικά δεν θα έχουν μετάφραση. Γίνεται μετάδοση μέσω διαδικτύου της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση για το αντίθετο, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των, των πρακτικών της προηγούμενης συνεδριάσεως του Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα εγκριθούν τα πρακτικά. Τρίτο θέμα. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι δεν έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος, άρα προχωράμε πολύ γρήγορα σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο θέμα στην σημερινή μας ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση της πειρατείας στον κόλπο της Γουινέας. Θα καλωσορίσω τους δύο σημερινούς ομιλητές μας, τον κύριο Βάντερ Μέρχετ της Μονάδας για τη Σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΔΕΦΚΟ και τον κύριο Ντόιλ, ε, επικεφαλής του Τμήματος Δυτικής Αφρικής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. No, okay. Uh, Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει το πρόβλημα της πειρατείας ε, μιλάμε κυρίως για αποστολές CSDP στο κέρας της Αφρικής, συνήθως. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τον κόλπο της Γουινέας. Χωρίς περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Βάντερ Μέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για την δραστηριότητά μας στη Δυτική Αφρική. Είναι τιμή μου που παίρνω για πρώτη φορά το λόγο στον χώρο αυτό. Θέλω να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι σύμφωνα με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει υλοποιηθεί ένα μέσο σταθερότητας και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και μέσα σε αυτή την προτεραιότητα υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την καταπολέμηση και την υποστήριξη κρίσιμων υποδομών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ασχοληθήκαμε με την Δυτική Αφρική κυρίως επειδή σημειώνουμε ότι οι δραστηριότητες μετακινούνται από την Ανατολική προς τη Δυτική Αφρική. Παρά τα αυτά υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά το ότι στη Δυτική το, τη Δυτική Αφρική ή τέλο πάντων τα πελάγη γύρω από τη Δυτική Αφρική στον κόλπο της Γουινέας οι δραστηριότητες έχουν σχέση ε, με πειρατεία που αφορά την κλοπή πετρελαίου. Αυτή είναι η διαφορά αν λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες ε, περιοχές. Μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμή έχουμε διαπιστώσει 98 περιπτώσεις, κυρίως ε, προελεύσεως Νιγηρίας, που έχουν ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Οπότε, είχαμε τον Ιούνιο μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο Γιαουντέ, όπου οι ηγέτες κεντρικής και δυτικής Αφρικής να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο για την αντιμετώπιση της πειρατείας. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί υποστηρίζει ουσιαστικά τη δουλειά μας. Θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκής πολιτική υποστήριξη σε αυτό που επιδιώκουμε σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους μας. Και κυρίως αφού διαβάσαμε τις δηλώσεις που έγιναν με αυτή την ευκαιρία, διαπιστώνουμε ότι οι δραστηριότητες της ανατολικής πλευράς κυρίως ε, σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς του Τζιμπουτί εφαρμόζονται στην ε, περίπτωση της Δυτικής Αφρικής. Αυτό το οποίο κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που προσπαθεί να συνδέσει αυτή την πολιτική διαδικασία που μόλις περιέγραψα με ένα πρόγραμμα που ονομάζεται προστασία των κρίσιμων θαλασσίων οδών στον κόλπο της Γουινέας. Ένα ε, πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες όπου ε, μία κοινοπραξία που καθοδηγείται από ένα κράτος μέλος σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους προσπαθεί να ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η πειρατεία. Και ε, η δουλειά μας ε, έχει, αποτελείται από τέσσερα μέρη. Πρώτον, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους εταίρους μας για, σε δραστηριότητες αντιμετώπισης κρίσεων. Δεύτερον, να ενισχύσουμε τα νομικά πλαίσια ώστε να υπάρξει και η απαραίτητη νομική διαδικασία ώστε οι συλληφθέντες να αντιμετωπίζονται με βάση τις υποχρεώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τέλος, μια, ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών το οποίο δημιουργείται ώστε οι ίδιες οι χώρες να μπορούν ε, με κάποιο τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους εάν ε, υποψιάζονται ότι υπάρχουν πλοία ή δραστηριότητα που, δραστηριότητες που τους δημιουργούν υποψίες. Αυτό ε, καταστάθηκε στο Καμερούν. Και βεβαίως η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειακών δραστηριοτήτων είναι και αυτή κομμάτι της δουλειάς μας. Ε, κύριε Πρόεδρε, το έργο αυτό μπορεί να πετύχει μόνο με την πλήρη υποστήριξη των χωρών εταίρων. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με τις, με αρχές του Μπενίν, του Τόγκο, του, της, της ε, Νιγηρίας ε, και της Δαχομέης που συμμετέχουν. Προσπαθούμε μέσω της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας μας και ε, να πετύχουμε συνεργασία ε, από την κυβέρνηση του Γκαμπών και της ε, Γουινέας του Ισημερινού. Είναι σημαντικό να υπάρξει εθνική συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό προσπαθούμε να θεσπίσουμε εθνικούς εθνικούς ανταποκριτές στα μέρη αυτά με τους οποίους θα είμαστε σε επαφή. Μετά από ένα διάστημα μηνών ημινών ε, υπάρχουν και τα πρώτα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Όμως είναι σαφές ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι προσπάθειές μας για να μπορέσει πραγματικά να γίνει δουλειά. Για να είμαστε ειλικρινείς, το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Πρώτον, διότι το αντικείμενο είναι αμφιλεγόμενο, είναι δύσκολο αντικείμενο. Δεύτερον, εξακολουθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να ψάχνουμε για τους ε, κατάλληλους εταίρους τις χώρες με τις οποίες θέλουμε να δουλέψουμε. Τέλος, ε, η εμπειρία μας από άλλα θαλάσσια προγράμματα είτε στο κέρας της Αφρικής είτε και αλλού θα μεταφερθεί φυσικά στο πρόγραμμα αυτό. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας αναφέρω ότι σκοπεύουμε να προωθήσουμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας στον Ινδικό ωκεανό και αυτό πιθανόν να αποτελέσει αντικείμενο κάποιες άλλες συζήτησης στο μέλλον με την υποεπιτροπή σας. Αυτά είχα να πω εν συντομία σχετικά με το πρόγραμμά μας στη Δυτική Αφρική Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι από την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα σας ε, πούν περισσότερα για αυτά που γίνονται στον τομέα αυτό. Επαναλαμβάνω όμως για μία ακόμα φορά ότι το όλο θέμα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών αποτελεί σημαντικό σκέλος της δουλειάς μας ε, και επιδιώκουμε σταθερότητα. Ελπίζουμε επίσης ότι θα επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων μας στην περιοχή αυτή του κόσμου. Thank you very much, Mr. Van der Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαντενμέρ και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο Ντόλ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τη συνάδελφό μου την κυρία Ντέιβις εργαζόμαστε στην υπηρεσία ε, Δυτικής Αφρικής ε, της υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης που όπως γνωρίζετε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες κυρίως όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρόκειται λοιπόν για μία, για μία σειρά νέων πρωτοβουλειών που ανελήφθησαν τους ε, τελευταίους μήνες. Ο συνάδελφός μου από την ΤΕΦΚΟ παρουσίασε το πρόγραμμα Gringo και την κατάσταση που αφορά ε, στο τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Επίσης ε, θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν όλο και περισσότερες επιθέσεις πειρατών στην περιοχή αυτή, Γκάνα, ε, η σημερινός ε, νέου γουινέα κατ' ουσίαν ε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των επιθέσεων και ο αριθμός των ναυτικών που δέχτηκαν επιθέσεις ήταν 966 το 12 σε σχέση με 851 στον κόλπο του Αίντεν. Η Νιγηρία βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά κατ' ουσίαν το πρόβλημα μεταφέρεται και μεταδίδεται και προς δεξιά και προς βοράν και προς νότον. Και αυτά δεν αφορούν μόνο την πειρατεία, αλλά αφορούν και τις συναφείς εγκληματικές δράσεις που πλήττουν την περιοχή. Όλα αυτά οφείλονται εν μέρη στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται ανάμεσα στη Λατινική και την Αμερική ε, σε αυτή την ε, μεταφορά ε, ναρκωτικών, ε, όπλων, ε, διακίνησης ανθρώπων, ναρκωτικά τα είπαμε αυτά. η πρόθεση λοιπόν είναι να αντιμετωπιστούν από κοινού όλα αυτά τα προβλήματα και κυρίως στο σύνολο της δυτικής ακτής της, της Αφρικής από την Σενεγάλη μέχρι την Αγγόλα και από, μέχρι και το πράσινο ακροτήρι. Τα θέματα βέβαια που συζητάμε δεν είναι τα ίδια όπως ακριβώς το κέρας της Αφρικής. Γιατί στο κέρας της Αφρικής βρισκόμαστε σε διεθνή ύδατα. Στην Δυτική Αφρική είμαστε μέσα σε ε, που εμπίπτουν στην επικράτεια συγκεκριμένων χωρών και με χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμφωνίες όπως με την Ιγυρία ή με τον Μπενίν. Η ε, προσπάθεια λοιπόν που χρειάζεται είναι τελείως διαφορετική από αυτήν ε, που χρειάζεται για το της Αφρικής και τη Σομαλία. Είναι περισσότερο θέμα συντονισμού, ανταλλαγής ε, πληροφοριών, υποδομής και αναγκαστικά πρέπει να προσέξουμε και τον εξοπλισμό. Όμως το θέμα δεν είναι ε, να τοποθετήσουμε κάποιους φρουρούς ε, μακριά από τις ακτές και να θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό λύσαμε το πρόβλημα. Η δική μας η προσέγγιση είναι η εξής. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που προτείνουν οι δύο περιφερειακές οργανώσεις και οι συναντήσεις τους που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο όπου συναντήθηκαν οι αρχηγοί των κρατών που συζητάμε και κατέληξαν σε μια κοινή προσέγγιση, σε ένα είδος στρατηγική ε, έναν κώδικα συμπεριφοράς, ε, τον οποίο πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά το γεγονός ότι οι δυνατότητες ε, είναι τελείως διαφορετικές όσον αφορά τις διάφορες χώρες. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ακόμα και αν κάποιες από τις χώρες αυτές επιθυμούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, δεν έχουν πολλές δυνατότητες. Βέβαια έλαβε χώρα αυτή η συνάντηση κορυφής, καθορίστηκαν πολιτικές και αυτό είναι ένα νέο μήνυμα που θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Επίσης θέλουμε να δουλέψουμε πάνω στην αρχή ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από την άλλη πλευρά της Αφρικής και ε, η πρόληψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα γιατί αν καθυστερήσουμε θα μας κοστίσει ε, πολύ περισσότερο. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να δράσουμε πριν προκληθούν περαιτέρω ζημιές. Ο στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο εξής. Θέλουμε κατά κύριο λόγο να επεξεργαστούμε μια στρατηγική από κοινού με τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, όχι μόνο με την ΤΕΦΚΟ, αλλά και με άλλες γενικές διευθύνσεις Επιτροπής, αλίας, εσωτερικών υποθέσεων, ε, μεταφορών, την πρώην μεταφορών, το περιβάλλον και πολλές άλλες γενικές ε, διευθύνσεις. Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία γίνεται της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Θεσμών συμπεριλαμβανομένου και του ε, Ταμείου Ανάπτυξης, του Εργαλείου για τη Σταθερότητα και πολλά άλλα. Ε, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο ε, θα απευθυντούμε και στην ομάδα εργασίας για την Αφρική του Συμβουλίου να το καλέσουμε να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη. Είχαμε κάποιες συναντήσεις με τα κράτη-μέλη και συζητήσαμε για θέματα αρχής. Καταλήξαμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχουν επικαλύψεις γιατί τελικά στον κόλπο της Γουινέας θα υπάρχει μια στρατηγική που δεν θα είναι η στρατηγική της Επιτροπής και κάποιων άλλων κρατών αλλά θα είναι μια αμυγής ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος λοιπόν είναι, όπως σας είπα, να αντιαστροπίσουμε όλα τα μέσα που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των προβλημάτων, όχι μόνο την πειρατεία που και αυτή δεν είναι εύκολο θέμα, να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα την εγκληματικότητα. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτά πρέπει να γίνουν κατά κύριο λόγο στην ξηρά και όχι στη θάλασσα, γιατί από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε βάθος, γιατί εδώ είναι θέμα θέματα ανάπτυξης και ασφάλειας. Όπως σας είπα λοιπόν, υπάρχει το στοιχείο του συντονισμού το οποίο θα είναι καθοριστική σημασίας και πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη ευελιξία με την έννοια πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι εφικτό για μας και για τα κράτη-μέλη πώς τα προβλήματα μετακινούνται με την έννοια ότι διάφορα κράτη ε, λαμβάνουν αντίμετρα και αυτό είναι γνωστό στην περίπτωση των ναρκωτικών. Ένα πρόβλημα μετακινείται σε άλλα πιο αδύναμα σημεία για να συνεχιστεί η μεταφορά ναρκωτικών. Άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην απάντησή μας. Επίσης πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Η βούληση δεν είναι παντού ίδια και αυτό απαιτεί ευελιξία εκ μέρους μας. Θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις της ε, συνθήκης της Λισαβόνας είναι ένα του στα χέρια μας για να μπορούμε να αξιολογήσουμε επιτόπου από κοινού τα κράτη-μέλη την πολιτική βούληση και για να δούμε επίσης ποιες είναι οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ποιες είναι οι προεκτάσεις τους και μήπως πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Η ευελιξία λοιπόν βρίσκεται στην πυρήνα του όλου θέματος. Και τέλος όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, παροχή πληροφοριών στις χώρες ε, στην Αφρική και μεταξύ μας βέβαια να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Όλα αυτά είναι υψής της σημασίας και αυτό αυτό που επιτιμούμε με τη στρατηγική μας είναι να υπάρχει μια γενική εικόνα, να υπάρχει σε γενικές γραμμές ανάληψη ευθυνών για όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, την κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ε, τα κρατημέλη και πολλούς άλλους. Και μετά να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα προγράμματα για συγκεκριμένα θέματα, τομείς και υποτομείς της περιοχής. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά αυτή είναι μια καινούρια προσέγγιση που θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα περιεκτικοί σε αυτά που κάνουμε. Ε, όλο αυτό το θέμα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το άλλο σκέλος είναι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα θέματα είναι τόσο σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους και είναι τώρα η στιγμή για ερωταπαντήσεις. Όπως είπα, έχουμε συζητήσει μια-δυο φορές το θέμα της επιχείρησης Αταλάντα και είναι σημαντικό να σας ρωτήσουμε τι διδάγματα αποκομίσατε από την επιχείρηση Αταλάντα. Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κόλπο της Γουινέας. γιατί η επιχείρηση Αταλάντα είναι ενδιαφέρουσα ως δική μας επιχείρηση, αλλά και όσον αφορά την συνεργασία με την επιχείρηση Ασπίδα των Ωκεανών του ΝΑΤΟ και συνεργασία και με τρίτες χώρες δηλαδή. Γι' αυτό θέλω να σας ε, θέσω αυτή την ερώτηση. Κυρία Κοπά, από την ομάδα των Σοσιαλιστών, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, εισήγηση. Σε αυτό το κοινοβούλιο είμαστε πολύ ευτυχείς και ε, συγχαρήκαμε την επιχείρηση Ταλάντα γιατί πιστεύουμε πως είναι ένα από τα σπουδαιότερα παραδείγματα της δυνατότητας που υπάρχει για μια επιχείρηση με συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Λίζικ ότι φυσικά πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από αυτή την επιχείρηση και επίσης θα ήθελα να έχω τα σχόλιά σας στο σημείο αυτό. Ταυτόχρονα ενώ περιορίζεται η πειρατεία στη Σομαλία, βλέπουμε να αυξάνονται επικίνδυνα οι επιθέσεις στην άλλη μεριά της Αφρικής, στον κόλπο της ε, Γουινέας. Εν γέννη, οι πειρατείες μειώθηκαν στο πρώτο ήμιση του 2013, αλλά σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, στον κόλπο της Γουινέας γίνανε επιθέσεις σε διάφορα είδη πλοίων, όπου βασικός στόχος των επιθέσεων ήταν η σύλληψη ομήρων. Ένα άλλο ανησυχητικό θέμα είναι ότι τα περιστατικά, τα πειρατικά δεν αναφέρονται έγκαιρα και αυτό δείχνει το χαμηλό βαθμό προετοιμασίας των τοπικών αρχών. Επίσης δείχνει ότι τα θύματα ε, δεν γνώριζαν τους, τις νέες επικίνδυνες περιοχές σαφές ότι είναι ότι οι ηγέτες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα υπεύθυνο σώμα που θα είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση της πειρατείας στον κόλπο της Γουινέας και η κρίση, το πρόγραμμα μάλλον για τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον κόλπο της Γουινέας μπορεί να βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια στις δυτικές ακτές της Αφρικής. Τώρα, συγκεκριμένη ερώτηση προς την Κομισιόν καταρχήν. Μπορούμε να γνωρίζουμε ποιε είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που προετοιμάζονται από το πρόγραμμα Gringo και έπειτα για, το, για την εξωτερική υπηρεσία δράσης για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, πιστεύετε ποιες θα, ποιοι θα είναι οι άξονες για μια ε, στεναρή πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας. Επίσης προβλέπετε μια συμμετοχή πολιτών πολιτικής άμυνας από πλευράς της ΚΠΑ. Στο κόλπο της Γουινέας. Ευχαριστούμε κυρία Κοπά. Άλλος που θέλει να θέσει ερώτηση. Okay, so... Okay, let's, uh, let's start for... Όχι, οπότε ας ακούσουμε τον κύριο Βαντεμέρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τα διδάγματα που αποκομίσαμε, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι στη δική μας ορολογία, σε σχέση με την Δυτική Αφρική, εμείς εφαρμόζουμε αυτό που θα έλεγα απαλά μέτρα θα το ονόμαζα και θα σας εξηγήσω ποια είναι αυτά τα μέτρα. Αλλά το κύριο δίδαμα που αποκομίσαμε από την άλλη πλευρά της Αφρικής, από το κέρας της Αφρικής, τον κόλπο του Άντεν, είναι για να το πούμε με μια λέξη, είναι το να ε, παρέμβουμε νωρίς, η έγκαιρη παρέμβαση. Δηλαδή, όταν γίνονται γεγονότα, όπως βλέπουμε τώρα, η προληπτική προσέγγιση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ότι η ε, διορθωτική προσέγγιση. Είμαστε λοιπόν ήδη εκεί, παρόντες στη Δυτική Αφρική με τη βάση αυτής της προληπτικής ε, προετοιμασίας, αλλά επίσης, όπως είπα και νωρίτερα, σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε το πολιτικό βάρος από τους αρχηγούς των ίδιων των χωρών, που κατά τη γνώμη μου πολύ πιο έγκαιρα από ότι στην άλλη πλευρά της Αφρικής αναγνώρισαν την ανάγκη συνεργασίας για αυτά τα θέματα, διότι πρόκειται πραγματικά για απειλή, απειλή στην ανάπτυξή τους να τονίσω ακόμη μια φορά αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι μόνο με ενός συνδυασμού μέτρων ανάπτυξης και ασφάλειας μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Έπειτα, σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα για την πτυχή της ασφάλειας και το πρόγραμμα Grimco, Έχουμε τέσσερα στοιχεία τα οποία εφαρμόζουμε, τέσσερα στατικά μάλλον, τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι η συνιστόσα κατάρτισης, ε, θαλάσσιας κατάρτισης όπου προσπαθούμε ε, να έχουμε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα ανταπόκριση σε κρίσεις στις εν λόγω χώρες. Δηλαδή στις ε, χώρες ε, της παράκτησης της Δυτικής Αφρικής. Και κάτι το άλλο που μπορεί να είναι εντυπωσιακό για κάποιον που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το γεγονός ότι δεν μοιράζονται σχεδόν καμιά πληροφορία οι χώρες για ύποπτα σκάφη ή ύποπτες ενέργειες δραστηριότητες στις χώρες αυτές. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και έχουμε κάνει και αλλού είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα πληροφορικής μέσω του οποίου να μπορούν επιγραμμικά, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, να μοιράζονται τις πληροφορίες οι αρχές αυτών των χωρών. Πολύ σημαντική πτυχή γιατί ελπίζουμε πως με αυτό το εργαλείο θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Αλλά σαφώς η έλλειψη ε, εξοπλισμού σε αυτές τις χώρες είναι κάτι που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε καθώς και την πυρογνωμοσύνη που λείπει για τη δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος. Επίτα από την ανάλυση μας είναι σαφές πως υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά νομικά κενά στις χώρες αυτές για να μπορέσει να υπάρξει μια προηγμένη πολιτική κατά της πειρατείας αλλά και να υπάρχει εγγύηση για δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πειρατές που συλλαμβάνονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην εργασία μας. Και τέλος, όπως είπαμε και πριν, όπως ακούστηκε πριν, το θέμα εξαρτάται πάρα πολύ από την ε, περιφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν δύο ε, οργανισμοί, η ECOWAS και η ECAS. Και αυτοί που, αυτό που προσπαθούμε είναι να ε, οικοδομήσουμε τις δικές τους δυνατότητες και να ε, μπορέσουν να συνεργαστούν και μεταξύ τους. και προσπαθούμε βέβαια να δούμε και συνεργασία με το γραμματεία του Συμβουλίου Δυτικής Αφρικής ώστε να εμπλοκεί και εκείνη στην ε, δουλειά αυτή, στην ε, όλη αυτή προσπάθεια. χρησιμοποιούμε την ε, τεχνογνωσία των κρατών μελών, αλλά και προσπαθούμε να δούμε και τι έχουμε στη διάθεσή μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα όσα έχουμε κάνει αλλού υπό τα προγράμματα για τα οποία συζητάμε εδώ και που είναι αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαντερμίρα. Ο κύριος Ντόλ. Ναι, αυτό. Πρώτα νομίζω πως θα πρέπει να τονίσω πως η κρίση, το πρόγραμμα μάλλον περί ε, κρίσιμων θαλασσίων οδών είναι ένα πρόγραμμα 45 εκατομμυρίων ευρώ για τις χώρες της ε, Δυτικής Αφρικής που μόνο δύο όμω είναι στην, ε, στις ακτές της Δυτικής Αφρικής. Η στρατηγική για τον κόλπο της Γουινέας είναι μια πολύ πιο ευρία, ε, ένα πολύ πιο ευρύ εγχείρημα έτσι ώστε να υπάρξει συνοχή ανάμεσα στι διάφορε δραστηριότητε, Το Κρίμγκο είναι μόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται όχι μόνο από τα κράτη-μέλη αλλά και από άλλα μέσα βοήθειας από πλευράς της ε, Κομισιόν. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα δηλαδή. Αυτή η νέα στρατηγική είναι πολύ ευρύτερη από το εν λόγω πρόγραμμα το Κρίμγκο. Ε, για να απαντήσω για την ερώτησή σας για την Αταλάντα, ο συνάδελφος ήδη ανέφερε το θέμα της πρόληψης και ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία ε, και θεωρούμε πως υπάρχει ανάγκη να συμμετέχουν όχι μόνο τα κρατημέλη αλλά και τρίτες χώρες εδώ. Δεν θα υπάρχει τίποτα κλειστό εδώ φυσικά και έχουμε εμείς μια δική μας ευρωπαϊκή στρατηγική αλλά αυτή μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο συντονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και όπου θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ε, συντονισμού ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αντίκτυπο και η ΕΠΑ η ΕΠΑ είναι μέγας παίκτη εκεί ίσως η Αμερικανική ακτοφυλακή να έχει κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον ε, στην περιοχή Τώρα, ε, στην ενδοχώρα ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα που αφορά την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Αυτό υιοθετήθηκε στις αρχές του 2011 παρά το πραξικόπημα στο Μαλί και τα γεγονότα στην Γουινέα Μπισάου. Παραμένει ωστόσο η βασική στρατηγική βάση για τα όσα κάνουμε σε αυτό το μέρος του κόσμου και προσπαθούμε να το επεκτείνουμε στο Ινμπουργίνα Φάσο και στο Τσάντ σε μια πρώτη φάση και επίσης το εμβαθύνουμε, δηλαδή αναπτύσσουμε κάποια μέτρα πολιτικής ασφάλειας. Θα γίνει συζήτηση στην Πολιτική Επιτροπή και Πολιτική Ασφάλεια στις επόμενες ημέρες όσον αφορά το πεδίο επέκτασης αυτής της στρατηγικής. Το μήνυμα είναι ε, πόσο σημαντική είναι μια τέτοια σφαιρική ε, προσέγγιση όπου συμμετέχουν όλα τα κοινοτικά μέσα αλλά και τα διαθέσιμα μέσα της ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ε, όπως το τόνισε και ο επικεφαλή ε, της, δική μας αντιπροσωπείας στον Ήγηρα, αλλά και το, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεών μας στο Μαλί. Το θέμα των ομήρων Αυτός ήταν ο στόχος των πειρατών στην ε, Ανατολική Αφρική εδώ και αρκετό καιρό και ένας μέγας φόβος που έχουμε είναι ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί μια δημοφιλής δραστηριότητα και στην Δυτική Αφρική. Δεν έχει αρχίσει ακόμα και δεν έχει φτάσει ακόμα στη μέγεθος ή στην κλίμακα που έφτασε στην ανατολική πλευρά της Αφρικής και αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα νομίζω που φαίνεται πως η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Δεύτερον, όσον αφορά την γνώση των ε, ναυτιλιακών εταιριών σε σχέση με τις απειλές. Ε, εγώ νομίζω πως γνωρίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείε τις απειλές, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη οποιασδήποτε μορφής πραγματικής διακυβέρνησης σε αυτές τις χώρες, στις περισσότερες, ε, και υπάρχει και ένα μέγα μειονέκτημα όσον αφορά τα ασφαλιστικά κόστη, για να δηλώσουν δηλαδή οι ναυτιλιακές εταιρείε το τι συμβαίνει είναι ε, ενδυμική, ενδυμικό το πρόβλημα της υποαναφοράς των όσων γίνονται εκεί. Όσον αφορά τους, ναύτες που δέχτηκαν, τους ναυτικούς που δέχτηκαν επιθέσεις, μάλλον είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των ε, όσων έχουν δεχτεί επιθέσεις στην πραγματικότητα. Τώρα, η μελλοντική μας στρατηγική. Εμείς θεωρούμε πως αυτή εντάσσεται ε, εν γέννη στην ε, θαλάσσια μας στρατηγική. Ε, αλλά το είδος των δραστηριοτήτων που εξετάζουμε είναι καταρχήν ενημέρωση και συντονισμός, να δημιουργηθεί μια κοινή συνεννόηση ανάμεσα στις χώρες ε, της περιοχής, ανάμεσα στους δύο ή τρεις περιφερειακούς οργανισμούς, αν μετρήσουμε και την Επιτροπή του Κόλπου της Γουινέας, Δεύτερον, η δημιουργία θεσμών και εν γέννη δημιουργία δυνατοτήτων στις διάφορες χώρες, αλλά και εντός των ε, διαφόρων οργανισμών όπως ECOWAS στην Αμπούντα στην ε, Νιγηρία και ΕΚΑΣ στην ε, Κεντρική Αφρική. Έπειτα, αντιμετώπιση των αιτίων όλων αυτών. Υπάρχουν προγράμματα αλλά προσπαθούμε να στοχεύσουμε περισσότερο τις παράκτιες περιοχές όπου περιλαμβάνεται ένα στοιχείο αλευτικής πολιτικής και αλευτικών συμφωνιών. Επίσης, προσπαθούμε να καλύψουμε το θέμα της ε, υποαπασχόλησης και της ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα σε όλα, σε όλα τα κράτη της, τα παράκτια. Και επίσης προσπαθούμε να οικοδομήσουμε δομές συνεργασίας ανάμεσα σε όλες αυτές τις χώρες οι οποίες δεν έχουν νομοθεσία καταρχήν κατάλληλη, δεν έχουν δικαστικό σύστημα ούτε μια δικαστική αλυσίδα που να μπορεί να αντιμετωπίσει τους όσους συλληφθούν. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν διαρθρωτικό δομικό έργο που πρέπει να γίνει ανάμεσα στις χώρες, μέσα στην κάθε χώρα και ανάμεσα στους περιφερειακούς οργανισμούς τους ίδιους οποιοδήποτε είδος παραδοσιακής ανάπτυξης δραστηριότητας ανάμεσα ε, που μπορείτε μάλλον να φανταστείτε δεν μπορεί να ε, ε, σταθεί εκεί. Τώρα, η συμμετοχή της ΚΠΑ είναι παρόμοια με αυτό που κάνουμε στο Σαχέλ. Δημιουργία δυνατοτήτων για το στρατητικό και για το πολιτικό σκέλος, η διδημοποίηση διαφόρων, αδελφοποίηση μάλλον διαφόρων θεσμών για να στηρίξουμε τους θεσμούς εκεί, ίσως και η δημιουργία θεσμών αλλά και το είδος διευκόλυνσης όσον αφορά την ε, συλλογή ε, προσφορών για εξοπλισμό όπως όπως συλλέχθηκαν από την αποστολή στο Μαλί, την αίμα, όταν είδαμε το πρόβλημα ε, που υπήρχε με την έλλειψη εξοπλισμού για την εκπαίδευση των στατευμάτων εκεί και όπως είπα νωρίτερα στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα κουτί ή να, περιορίσουμε και όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για μια στρατηγική όπου να μπορεί να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότεροι να αντιμετωπίσουμε τα κενά και να μετά να καταρτήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μπορώ να πω ότι είναι βέβαιο ότι η Υποεπιτροπή μας θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις και ενδεχομένως θα μιλήσουμε και στο μέλλον για τα θέματα των συνεργασιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριοι. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα ε, το οποίο είναι σίγουρα ενδιαφέρον, ίσως και να προκαλέσει ενθουσιασμό. Περιμένω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των μελών. Θα μιλήσουμε για την πυραυλική άμυνα και την κατάστασή της. Έχουμε δύο ομιλητές. Ο ένας είναι ο κύριος Ρομπέτρο Ζάντρα, επικεφαλής του Τμήματος Άμυνας Καταβαλιστικών Πυράβλων του ΝΑΤΟ. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Νικολάη Κορτσούνοφ, ασκών καθήκοντα μονίμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Προσκαλέσαμε επίσης το Ινστιτούτο τον κύριο Φλάνς Κλέχικ από το Ινστιτούτο Μελετών του Ειρηνικού και λοιπά, αλλά θα σας ζητήσω εσείς να κλείσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε περισσότερο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζάντρα για να μας παρουσιάσει τα τεκτενόμενα, τα σχεδιαζόμενα και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα της ε, πυραυλικής άμυνας. Για να διευκρινίσουμε πόση ώρα για πόση ώρα μου δίνετε το λόγο. Συνήθως ε, δίνουμε το λόγο για 8 10 λεπτά στους ομιλητές και κατόπιν ακολουθούν ερωτήσεις και άρα μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Έχω την αμφιλεγόμενη χαρά να είμαι επικεφαλής ε, των πολιτικο-στρατιωτικών συζητήσεων του ΝΑΤΟ για το αντιπυραυλική άμυνα και τις συζητήσεις για το ίδιο θέμα με τη Ρωσία. Και αν ήθελα να ανακεφαλαιώσω με δύο λόγια το που βρισκόμαστε, μπορώ να πω τέσσερα ίσως πράγματα. Πρώτον, στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την ε, ανάπτυξη μέχρι τώρα θα μπορούσα, στο ΝΑΤΟ θα μπορούσα να πω καλά τα πάμε μέχρι τώρα. Η δουλειά του ΝΑΤΟ προχωρεί σε γενικές γραμμές ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όπως θα ξέρετε μετά την διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας του 2010, 18 μήνες αργότερα στο Σικάγο αποφασίστηκε, ανακοινώθηκε ότι το ΝΑΤΟ είναι η ενδιάμεση δυνατότητα, πράγμα που αποτελεί σημαντικό βήμα πρόοδου και επιχειρησιακά. Αυτή η ενδιάμεση δυνατότητα επίκεντρο έχει την προστασία με τα διαθέσιμα μέσα των των πληθυσμών και των εγκαταστάσεων κλπ. από πιθανές ε, επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων. Αυτό τι σημαίνει. Στην ουσία σημαίνει ότι παραδέχεται το ΝΑΤΟ ότι ότι η ενδιάμεση προσωρινή δυνατότητα δεν μπορεί να προστατεύσει τα πάντα από τα πάντα. Είναι ακόμα περιορισμένη. Ουσιαστικά Ε, σε συνδυάζεται με το, τις συσκευές αναχέτησης στη Μεσέγειο συμπεριλαμβανομένης και του ραντάρ, συμπεριλαμβανομένου και του ραντάρ της Τουρκίας και μετά υπάρχει το σκέλος ε, δι, ε, και έλεγχος που υπάρχει στη Γερμανία. Τώρα το δεύτερο προς τα που κατευθύνεται το ΝΑΤΟ και πότε θα φτάσει εκεί που πηγαίνει στόχος, όπως γνωρίζετε, της ε, επιχείρησης του ΝΑΤΟ είναι να καλυφθούν όλοι οι πληθυσμοί, τα εδάφη και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό θα χρειαστεί χρόνια, ε, ίσως ε, την υπόλοιπη δεκαετία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπουν τρεις φάσεις. Έχουμε τις θέσεις EPAA 1, 2 και 3, οι οποίες σκοπός είναι να ολοκληρωθούν εντός του 2000, μέχρι το 2018, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η τρίτη φάση, αλλά περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν ώστε η συνολική δυνατότητα να ενισχυθεί ποια είναι τα ε, οι επόμενες επιδιώξεις αφού έγιναν οι ανακοινώσεις της ε, Λισαβόνας και μετά του Σικάγο. Οι επόμενες επιδιώξεις θα είναι να φτάσουμε την, ε, την κατάσταση όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα μπορούν να ανακηρύξουν αρχική, επιχειρησιακή δυνατότητα και κατόπιν πλήρη. AFC και ε, ROC. Τώρα πότε το IOC και το FOC αυτή τη στιγμή συζητώνται, δεν ξέρουμε πότε θα εκπληρωθούν. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις αυτές. Οπωσδήποτε οι δυνατότητες, αλλά εξίσου δυνατό, ε, σημαντικό είναι η, τα στοιχεία της, του ελέγχου και διοίκησης στο ευρύτερο στρατιωτικό πλαίσιο, που και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τρίτο στοιχείο. Η εθνική συνεισφορά προς την ε, αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ η κοινά χρηματοδοτούμενη, ε, το κοινό χρηματοδοτούμενο σκέλος του ΝΑΤΟ αφορά τον έλεγχο και τη διοίκηση ε, που χρηματοδοτείται και από τους 28 συμμάχους. Οι, αναστολ, οι αναχαιτιστές και οι sensors χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή χρηματοδότηση και μετά υπάρχει χρηματοδότηση από τα κράτη ή από συγκεκριμένα προγράμματα. Επιπλέον, όπως είπα πριν, υπάρχουν, θα ήταν χρήσιμες οι επιπλέον εθελοντικές εθνικές συνεισφορές για να αυξηθούν οι δυνατότητες. Ξέρουμε ότι οι σύμμαχοι εξετάζουν ενδεχόμενο συνεισφοράς. Αναμένουμε αυτές οι επιπλέον συνεισφορές να γίνουν βαθμιαία και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει δυνατότητα για πολυμερή συνεργασία. Τώρα το τελευταίο σημείο μου, το τέταρτο και τελευταίο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ και ενδεχομένως και το πιο δύσκολο, αλλά έχω εδώ έναν διακεκριμένο συνάδελφο που θα μπορέσει να επεκταθεί, είναι η συνεργασία με τη Ρωσία. Στη Λισαβόνα το 2010 ουσιαστικά και αυτό φαίνεται και από την δήλωση του κειμένου της Λισαβόνας. Υπάρχει ένας διπλός σκοπός. Αφενός, λήφθη απόφαση να ε, αναπτυχθεί η ικανότητα του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα διατυπώθηκε μέσω μιας προσφοράς που έκανε η, το ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία να συνεργαστούμε για την ε, πυραυλική άμυνα. Άρα, ο διπλός αυτός στόχος δεν μοιάζει ότι επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή. Το έργο του ΝΑΤΟ προχωρεί, όμως η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην πυραυλική άμυνα όχι. Όπως είπα είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας εργασίας, συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας ε, για την πυραυλική άμυνα και πρέπει να πούμε ότι το 2013 ε, ήταν απογοητευτική χρονιά για μένα και δεν είμαι ο μόνος γιατί, επειδή είχαμε διάφορες εντολές που προήρθαν από το, τη διασκεψη κορφή κορφής ΝΑΤΟ-Ρωσίας ε, του 2010 για να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο μελλοντική συνεργασίας. Οι εργασίες αυτές έχουν καθυστερήσει και έχουν πέσει στα στασιμότητα. Και η δεύτερη εντολή ήταν να, να, να επαναλάβουμε τη συνεργασία TMD. Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι την Άνοιξη στη Γερμανία και σκοπεύαμε να συνεχίσουμε αλλά και εδώ υπάρχει στασιμότητα. Έχουν γίνει από πλευράς ΝΑΤΟ επιπλέον προτάσεις στο Σικάγο. Δεν είχε γίνει ε, τότε διάσκεψη κορυφής NRC με τη Ρωσία δηλαδή και είχε προς προσφερθεί τότε συνεργασία για την πυραυλική άμυνα και ένα καθεστώς διαφάνειας στην πυραυλική άμυνα προς, με τη Ρωσία. Όλες αυτές οι δυνατότητες δεν έχουν διερευνηθεί στο βαθμό λεπτομέρειας που θα ήθελα εγώ. Έγιναν κάποιες αρχικές συζητήσεις, αλλά όχι κάτι το προχωρημένο. Με δύο λόγια, δηλαδή τίποτα δεν προχωρήσουν το με αυτό. Θεωρώ πρόεδρο της ομάδας ε, σε στασιμότητα και ελπίζουμε ότι θα επανέλθει και θα βρούμε ένα τρόπο κοινό να προχωρήσουμε και να ξεπεράσουμε τις θεμελιώδεις διαφορές. διαφορές. Οι θεμελιώδεις διαφορές που έχουμε αφορούν τη συζήτηση για ένα κοινό σύστημα ή ένα χωριστό σύστημα που θα συντονίζεται η Ρωσία έχει ζητήσει νομικές διαβεβαιώσεις και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν προχωρούμε. Τρία χρόνια τώρα. Ε, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε πρόοδο. Τη φάση αυτή δεν είμαι ιδιαίτερο αισιόδοξο, παρότι είμαι αισιόδοξο άνθρωπος. Δεν είμαι ιδιαίτερο αισιόδοξο. Γνωρίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν δεν υπάρξει διμερής συμφωνία για το πώς θα προχωρήσει μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία. Δηλαδή, αυτό είναι θεμελιώδος. Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας μπορεί να προσφέρει πολλά, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την διμερή στρατηγική σχέση. Στο σημείο αυτό θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αργότερα θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση. Κύριε Πρέσβη. Όπως ε, γνωρίζουμε υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα με το πρόγραμμα αυτό ανάμεσα στους πολιτικούς της Ρωσίας και την κυβέρνηση. Ε, πάρα πολλοί Ρώσοι πάρα πολλά στελέχη στη Ρωσία είναι επιφυλακτικά. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας εκφράσετε και εσείς την άποψη της Ρωσίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και κοντά στον Ρόμπερτ γιατί συνεργαζόμαστε ε, στενά. Συμφωνώ Ρόμπερτ με αυτά που είπατε σχετικά με το ότι πράγματι η Ρωσία θέλει τη συνεργασία. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση πραγμάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σας υπενθυμίσω το Φόρουμ των Βρυξελών του Μαρτίου του 2010 Ο κύριος Ράσμουσεν τότε πρότεινε να υπάρχει ε, ένα ανώτατο επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά την αντιπυραυλική άμυνα. Αυτό ε, σημαίνει και σήμανε ότι συνεργαστήκαμε να υπάρχει ένα ανώτατο όριο αυτό κατ' ουσίαν σημαίνει βέβαια ότι ε, θα πρέπει να μοιραζόμαστε και τα ωφέλη και το κόστος. Έτσι λοιπόν είχαμε την δήλωση τελικά του Συμβουλίου Ρωσίας-ΝΑΤΟ σχετικά με την ε, αντιπυραυλική άμυνα. Ο στόχος, όπως είπε και ο Ρόμπερτ, ήταν να καθοριστεί ένα πλαίσιο για την αντιπυραυλική άμυνα και να υπάρχει συνεργασία. Δυστυχώς όμως οι συζητήσεις ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες κατέδειξαν ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ο κ. Μεδιέντεφ τότε πρότεινε να υπάρχει ένα σύστημα που να ε, προστατεύει τους πληθυσμούς μας ε, από βαλιστικές επιθέσεις εκτός της Ευρώπης. Ε, θα είχαμε μία πυραυλική ομπρέλα όπου η Ρωσία και το ΝΑΤΟ θα ήταν ισότιμοι εταίροι. Από την άλλη βέβαια ε, υπήρχε το άρθρο 5 της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ που αναφέρεται ότι οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να βασίζεται μόνο σε δύο ε, ξεχωριστά αλλά συντονισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν σημαίνει να υπάρχουν δύο μπρέλες ε, που να λειτουργούν παράλληλα. Αυτή λοιπόν η παραδοχή των δύο διαφορετικών συστημάτων όμως δεν έλυνε τα βασικά προβλήματα της Ρωσίας. Δηλαδή υπήρχε ανησυχία ότι το σύστημα που θα ε, εισήγεται στην Ευρώπη από τις Ηνωμένε Πολιτείες ή κάθετος ΝΑΤΟ ε, και τις δύο δηλαδή αυτές δυνάμεις θα ήταν κατά της Ρωσίας. Μετά Τη συνάντηση στη Λισαβόνα οι συζητήσεις ε, πλέον παρουσίασαν στασιμότητα. Μπορέσαμε όμως ε, να κάνουμε μια ε, προσωμείωση το Μάρτιο του 2012 και εστιάσαμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα εδαφικά στοιχεία πυραυλικής άμυνας και από εκεί φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα της ε, πυραυλικής άμυνας αυξάνεται και με το αυξανόμενο επίπεδο επιχειρήσεων. Συγκρίναμε λοιπόν τα αποτελέσματα του μοντέλου του του ΝΑΤΟ με δύο συντονισμένα συστήματα πυραυλικά. Όλα αυτά τα συγκρίναμε και με τα ρωσικά συστήματα για να καταλήξουμε ίσως σε ένα κοινό σύστημα και φάνηκε ότι το κοινό σύστημα θα ήταν το καλύτερο. Όταν όμως προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα συντάξουμε σε μια συγκεκριμένη έκθεση μετά τη δράση. Ορισμένα ε, κράτη-μέλη διαφώνησαν γιατί προφανώς ε, δεν ήθελαν να ενταχθούν σε αυτή τη βαλιστική εικόνα. Κατόπιν τούτου οι συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας όπως είπε και ο Ρομπέρτο, οι συζητήσεις ε, διεκόπησαν. Δεν υπήρξε πρόοδος ε, και δεν υπάρχει πρόοδος για ένα περίπου χρόνο. Η βασική απόφαση της Λισαβόνας να υπάρχει κοινή ανάλυση ενός πλαισίου για τη συνεργασία, αυτή εφαρμόστηκε και οι ε, προπτικές ε, όμως για να μας ειλικρινείς είναι αρνητικές. Ε, αυτό είναι το ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που κάνει λόγο για την συνεργασία. Εμείς θελήσαμε το θέμα της πυραυλικής άμυνας να το εντάξουμε στην καθημερινή, στις καθημερινές συζητήσεις, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και εδώ προβάλλει κάτι άλλο. Δηλαδή όλοι και, όλο και περισσότεροι αγωνιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να αποτελούν κίνδυνο για τις στρατηγικές δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες τόσο για την Ευρώπη όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν σχέσεις ε, υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στον ε, στρατηγικό επιθετικό βραχίωνα και αυτόν τον αμυντικό βραχίωνα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν ένα μέρος προσπαθήσει να αυξήσει την αμυντική του ικανότητα με αυτόν τον τρόπο μειώνει τις, ε, ε, πυραυλι... τις πυρηνικές εκφοβιστικές δυνατότητες της άλλης πλευράς και καλείται η άλλη πλευρά να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Αυτό όμως προκαλεί αστάθεια και κατόπιν τούτου υπάρχει λιγότερη ασφάλεια και λιγότερη προβλεψιμότητα για όλους. Πόσο μάλλον για τα οπλοστάσια. Δεν είμαστε οι μόνοι που ανησυχούμε. Υπάρχουν και άλλες χώρες που αναφέρουν ότι και η Κίνα εξυγχρονίζει και επεκτείνει το ε, πυρηνικό της ε, οπλοστάσιο για να ε, ανταποκριθεί στην επέκταση της πυραυλικής άμυνας και αυτό οδηγεί στο να αντιδράσουν και άλλες δυνάμεις και δημιουργείται μια επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Αλλά ας επανέλθουμε στην Ευρώπη. Στη Μόσχα η συνδιάσκεψη για την ασφάλεια ε, φέτος και πέρυσι υποβάλαμε υπολογισμούς που δείχνουν ότι η πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ αποτελούν κίνδυνο για τις ρωσικές δυνάμεις. Η τέταρτη φάση για την πυραυλική άμυνα στην Ευρώπη ε, δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες μας και υπάρχουν τρία θέματα που αποτελούν κίνδυνο για μας. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο. Η, τα σκάφη με αναχαιτιστικές ε, συσκευές ε, και συστήματα και αυτά αποτελούν πρόβλημα για μας. Εδώ λοιπόν ε, θα ήθελα να σας επισημάνω και τη συμφωνία που έγινε με το Ιράν για τα πυρηνικά όπλα. Η απειλή από το Ιράν αναφέρθηκε επανειλημμένα γιατί θα πρέπει στην Ευρώπη να αναπτυχθούν βαλιστικά αμυντικά συστήματα. Ο κ. Λαυρόφ είπε ότι ο βασικός λόγος ε, γιατί να υπάρχουν ε, ε, αυτά τα αισθήματα στην Ευρώπη υποτίθεται είναι το, η απειλή από το Ιράν. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή και εξακολουθεί να υπάρχουν τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, η Ρωσία θα συνεχίσει να ανησυχεί για το πού ακριβώς μπορεί να κατευθυνθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να έχει κανείς μεγάλη φαντασία για να μιλάει ε, για απειλή ε, στην Ευρώπη από τη Βόρειο Κορέα. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς ε, και να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο, ο κύριος Ομπάμα στην ομιλία του στην Πράγα το 2009 είπε η εξάλληψη της απειλής από το Ιράν θα μετακινήσει ε, την ε, πυραυλική άμυνα στην Ευρώπη. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ε, ανησυχούν για την στρατηγική που ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικέ δυνάμεις. Από την άλλη πρέπει να πω ότι δεν έχουμε δει να υπάρχει μέχρι τώρα μια απόδειξη ε, που να δείχνει ότι κάνουμε λάθος. Κάτσε άλλο. Ανταυτού το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν με την προσέγγιση τους, όπως ε, πριν από λίγο είπε και ο Ρόμπερτ. Όμως όσον αφορά την τελική λύση για την πυραυλική άμυνα, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη ε, για την Ρωσία να καταστήσει σαφές ότι οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν θα υπονομεύσουν τις δυνατότητες ε, αποτροπής ε, που, και εκφοβισμού που διαθέτει η Ρωσία. Υπάρχει ένας δεδηλωμένος στόχος που είναι η πρόληψη απέναντι σε ε, πυράβλους που θα μπορούσαν να προέρχονται ε, από χώρους εκτόξευσης εκτός Ευρώπης. Έχοντας κατά νου ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αυτά τα συστήματα τα αντιπυραυλικά θα πρέπει να έχουμε ε, την, κατά νου το σύνολο της Ευρώπης όχι μόνο τις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι, δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι λοιπόν η εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας που ισχύει για όλα τα κράτη, σε κάτι στο οποίο έχουν δεσμευτεί ε, όλα τα κράτη. Νομίζω αυτή η αρχή είναι σημαντικότερη από ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, ευρωβουλευτές. Κυρία Κοπά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγησή σας. Ε, σίγουρα δεν είναι εύκολο το θέμα ε, αυτό για να συζητηθεί τώρα όσον αφορά την ασπίδα, την αντιπυραυλική. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Κοτσούνοφ. Εμείς παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις μετά από την απόφαση σε σχέση με το Ιράν σε σχέση με το ότι δεν, ποτέ, δεν υπάρχει πλέον απειλή από το Ιράν και άρα ότι ίσως και ολόκληρο αυτό το project είναι άχρηστο. Μήπως μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερα. Δεν νομίζετε πως είναι κάπως νωρίς για να πει κανείς ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από το Ιράν. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή τη συμφωνία και είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά πιστεύω πως χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνος για να δούμε αν όλες οι ρήτρες της συμφωνίας ε, θα εφαρμοστούν. Ε, φοβούμε λοιπόν πως η Ρωσία λίγο βιαστικά ε, ασπάστηκε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να έχω την αντίδρασή σας λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κόντρακ. Thank you. I'd like to... Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το θέμα Ρωσία-ΝΑΤΟ και τη συνεργασία για την ε, αντιπυραυλική ασπίδα. Καταρχήν υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, αντιπυρευλικές άμυνες. Το ιδέα αρχικά ήταν να υπάρχει μία κοινή και στην παράγραφο 5 και εσείς κύριε Κοτώνοφ αναφερθήκατε στους λόγους της ύπαρξης των δύο χωριστών αντί για μία. Ναι, ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγος, αυτή είναι η λόγια, όχι. Ε, εγώ θέλω να θέσω την εξής ερώτηση όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας. Κατανοώ ότι αν υπάρξει μία ενιαία κοινή σπίδα θα υπάρξει μεταφορά ε, αμερικανικής τεχνολογίας προς τους Ρώσους και καταλαβαίνω τους λόγους των Αμερικανών που δεν το επιθυμούν. Η παράγραφος, πέμπτη παράγραφος είναι όντως λοιπόν ο λόγος και έπειτα υπάρχει και ένα θέμα νομικών και πολιτικών εγγύσεων. Ο, δηλαδή, η αντιπυραυλική άμυνα περισσότερο προορίζεται στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει ζητήσει νομικές εγγυήσεις και το ΝΑΤΟ δεν έχει δώσει μόνο πολιτική φύσης εγγύησης. Μπορείτε να το σχολιάσετε και από την πλευρά του ΝΑΤΟ αυτό, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Στέρκου που είναι εισηγητής μας για την έκθεση που τώρα αρχίζουμε να επεξεργαζόμαστε για τις πολιτικές και στρατηγικές επιπτώσεις της αντιπυροευλικής ε, ασπίδας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω για το ίδιο θέμα, όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια. Δεν κατάλαβα απόλυτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τώρα στις πραγματεύσεις, γιατί οι δύο πλευρές ε, φαίνονται να είναι εξαιρετικά πρόθυμες να συνεργαστούν. Ποια είναι τα πραγματικά συγκεκριμένα προβλήματα των διαπραγματεύσεων και από την άλλη πλευρά τι λύσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν. Ο κ. Κοτονόφ είπε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Για παράδειγμα, τι συγκεκριμένε εγγυήσει εννοείται ότι θα θέλατε από την άλλη πλευρά. Ευχαριστούμε κύριε Τέρχοφ. Ο κύριος Ζάμκε που είναι Πολωνός, υφυπουργός άμυνας της Πολωνίας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους στους ε, φιλοκριτούς μας και για τη δυνατότητα να ακούσουμε διαφορετικές γνώμες ε, σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ καλή ιδέα. Ε, με αυτή τη βάση θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Το σημείο κίνησης αυτής της συζήτησης πρέπει να είναι μια αξιολόγηση των απειλών που υπάρχουν όχι μόνο σήμερα αλλά και που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ή να προκύψουν στο μέλλον. Εδώ λοιπόν η ερώτηση. Έχω την εντύπωση πως υπάρχουν διαφορά απόψεων, διαφορά, διαφορά Πώ Πώς ορίζεται αυτές τις απειλές που μπορεί να προκύψουν στον ορίζοντα σε κάποια χρόνια. Και αυτό το ερώτημα δεν γίνεται άνευ ε, αιτίας, γιατί παρατηρούμε μια πραγματικότητα η οποία διαρκώς αλλάζει. Βλέπουμε τι συμβαίνει στο Ιράν, στο Ιράκ. Όλα αυτά δείχνουν πως Όλα αυτά που νομίζαμε ε, ότι θα είναι απειλές πριν από ένα χρόνο δεν παραμένουν πάντοτε απειλές. Δεύτερο ερώτημα για τον πρέσβη της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτό αυτή την επιχειρηματολογία. Η λειτουργία μιας τέτοιας ασπίδας θα περιόριζε τις δυνατότητες της Ρωσίας. Γνωρίζουμε πως η Ρωσία έχει, πολύ μεγα, έχει μεγάλο δυναμικό ε, κρούσης Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε με λεπτομέρειες γιατί αντίθετα οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ λένε το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν είναι αυτός ο στόχος, ότι ο στόχος της ασπίδας δεν είναι το να επηρεαστεί η θέση της Ρωσίας. Τρίτη ερώτηση. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτή η ασπίδα έχει, αποτελείται από διάφορα επίπεδα αυτή η κοινή σπίδα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο τους βαλιστικούς πύραυλους ή πρέπει να έχει δυνατότητες να μπορέσει να αναχαιτήσει και πύραυλους που, πηγαίνουν, που ταξιδεύουν σε πιο χαμηλό επίπεδο και έχουν και πιο περιορισμένο βεληνικές. Ε, σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις σας. Ε, θα ήθελα σύντομα να σας συστηθώ. Είμαι νέο μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά προηγουμένω ήμουν μέρος του PA της, ε, του ΝΑΤΟ από την Κροατία. Ερώτησή μου λοιπόν απευθύνεται στον κύριο Κοτσούνοφ. Αναφέρατε στην τελευταίο κομμάτι της ε, εισήγησή σας τη σημασία του ΝΑΤΟ και ε, της των σχέσεων μάλλον ΝΑΤΟ-Ρωσίας ε, για χώρες εκτός νατο επειδή η χώρα μου είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μέσα στο ΝΑΤΟ προσπαθούμε να έχουμε στενές σχέσεις με αυτές τις χώρες, το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι πιστεύετε, πώς αυτό θα επηρέαζε την κατάσταση της ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προτείνω τώρα να πάρει το λόγο ο πρέσβης Κοντούνοφ για 5-6 λεπτά. Τόσες πολλές ερωτήσεις που δεν είναι εύκολο να τις σημειώσει κανείς, αλλά ας ξεκινήσω από την κυρία Κοπά που ρώτησε μήπως είναι πρόημο το συμπέρασμά μας, όπως είπε ο κύριος ο Υπουργός Λαυρόφ, για το ότι το, αν λύθηκε το ιρανικό πρόβλημα, οπότε δεν χρειάζεται η, πυραυλη, η πυραυλική άμυνα που κατασκευάζει το ΝΑΤΟ. Ναι, είναι πρόημο να πει κανείς κάτι τέτοιο, ωστόσο είναι η αρχή μιας τέτοιας διαδικασίας διαβουλεύσεων. Ε, αν δούμε Εάν υπάρχουν, ε, αν δούμε ότι αν, δεν αν θεωρήσουμε μάλλον ότι εάν δεν υπάρχουν η ε, απειλή, από το Ιράν, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος, ε, ναι, ε, ε, όντως δεν είναι, γιατί για την περιοχή του Ειρηνικού η Βόρεια Κορέα είναι η απειλή. Και έπειτα θα ήθελα να κάνω μια, ένα σχόλιο στρατηγικής ευθύσης από το χώρο των στατικικών μελετών ότι το Ιράν δεν θα έχει ICDM τουλάχιστον για 10 ακόμα χρόνια. Το σχόλιο αυτό αφορά την ερώτηση που εσείς ε, γύρατε. Το άρθρο 5 κατά πόσο εμείς οι Ρώσοι θεωρούμε πως αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο για το ΝΑΤΟ και για την ύπαρξη μάλλον ε, ε, μίας ενιαίας ε, αντιπυραυλικής άμυνας με το ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι πώς ερμηνεύει κανείς αυτό το άρθρο παιδί, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για μια συμφωνία 60 ετών. Εάν υπάρχουν ε, στρατεύματα χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και συμβάλλουν κάποιες από τις χώρες του ΝΑΤΟ οικονομικά αλλά και με υλικό ε, για αυτά τα στρατεύματα ώστε να παρέχουν ασφάλεια εκεί είναι αυτό θέμα εγγύησης ή όχι. Υπάρχουν και τέτοιου είδους ζητήματα και όσον αφορά τη μεταφορά ε, τεχνολογίας οι Αμερικανοί δεν νομίζω ότι επιθυμούν ιδιαίτερως να μεταφέρουν ε, τεχνολογία τους ε, ούτε και στους Ευρωπαίους. Είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα και εμείς κάνουμε τέτοια πρόταση να υπάρχει ένα μόνο ενιαίο πρόγραμμα, ένα ενιαίο σύστημα, όχι έχοντας την υπόψη μας το να πάρουμε την τεχνολογία των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί είναι πολύ καλοί στο να ε, Ε, καλύπτουν και να αποκτούν τις πληροφορίες που θέλουν, αλλά έχουμε και εμείς ένα δικό μας πολύ καλό ρωσικό σύστημα. Με τους Αμερικανούς θα μπορούσαμε, θέλουμε να συνεργαστούμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν ε, προβλέπαμε τίποτα τέτοιο, καμιά μεταφορά τεχνογνωσίας από τους Αμερικανούς εδώ. Αλλά νομίζω ίσως ο Ρομπέρτο θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Πολιτικές εγγυήσεις. Ε, βεβαίως οι πολιτικές εγγυήσεις ε, είναι σημαντικές αλλά ευμετάβλητες. Αν ερχόταν ας πούμε μια νέα κυβέρνηση στο Λευκό Οίκο, ο π.χ. ο Μακέιν ή κάποιος άλλος υποψήφιος μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Αυτό που έχουμε ως νομική εγγύηση μπορεί να καταστήσει τη σχέση μας σταθερή και βιώσιμη. τουλάχιστον για κάποιο ε, χρονικό διάστημα. Τώρα, τι είδους εγγυήσει ασφαλείας χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ευρύτατες εγγύησεις ασφαλείας ε, που θα είναι βαθύτερες ε, πέρα από το ότι το σύστημα αυτό δεν είναι μόνο για την Ρωσία. Θέλουμε συμφωνία στο επιχάρτου. Πόσες ε, δυνατότητες αναχέτησης χρειάζεται για να μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή από τον Νότο 100, 200 ε, συστήματα. Αλλά όταν βλέπουμε τι συγκεκριμένου χώρους τοποθεσίες και το σχεδιασμό αυτών στη Ρουμανία και την Πολωνία, έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Γιατί υποτίθεται πως το σύστημα αυτό θέλει να αντιμετωπίσει την νότια απειλή Και εμεί λέμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Άμυνα μαζί. Να τη σχεδιάσουμε. Αυτά είπε και ο Ράσμουσεν το 2010. Φτιάχνουμε μαζί, στηρίζουμε μαζί, ε, μοιραζόμαστε το κόστος μαζί, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις μετά έδειξαν πως ε, Ε, ε, έδειξαν ότι από την πλευρά του ΝΑΤΟ όλα αυτά εξελίχθηκαν προς άλλη κατεύθυνση. Uh, of course, threat assessment is, is very important, but uh, missile threats. Είναι σημαντικές, σημαντική η πύραυλη φυσικά, αλλά και στο πλαίσιο των χωρών του ΝΑΤΟ υπάρχουν διαφωνίες στον τομέα αυτό. Ε, και κατόπιν έχουμε το ερώτημα των Βαλκανίων και της Ρωσίας και ποιες είναι οι επιπτώσεις, πώς επηρεάζεται η Βαλκανική. Αν κατάλαβα καλά. Η Βαλκανική δεν είναι κοντά στη Ρωσία. Είναι μία από τις περιοχές Υπάρχουν χώρες που θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και άλλες χώρες όπως η Σερβία έχουν τις επιφυλάξεις τους. Από την άλλη πλευρά η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ο οποίος είπε ότι όλη η περιοχή θα πρέπει να ενσωματωθεί στις ατλαντικές δομές αν η Σερβία έχει επιφυλάξεις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψή τη. Ακόμα και από έναν τόσο ψηλό βαθμό αξιωματούχο όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας που ταυτόχρονα είναι πρόεδρος του Συμβουλίου ΝΑΤΟ Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάντρα, θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς σε κάποια από αυτά που είπε ο πρέσβης. Ναι, θα προσπαθήσω να το κλείσω και να απαντήσω σε κάποια σχόλια. Καταρχήν, έχει γίνει πολιτική δήλωση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ότι η πυραυλική άμυνα του νατο δεν στρέφεται κατά της ρωσίας και δεν θα συμβεί αυτό. όχι μόνο δεν, γίνεται, δεν ισχύει τώρα αλλά δεν θα ισχύσει. Αυτή η δέσμευση δόθηκε γραπτά από τους αρχηγούς κρατών ε, του ΝΑΤΟ. Παραδέχτηκαν ότι υπάρχει αίτημα για νομικές εγγυήσεις. Υποστηρίζω όμως ότι επειδή υπάρχει πολιτική δέσμευση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο από 28 κράτη, ήδη έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό καθησυχαστικό στοιχείο. Το πρώτο. Δεύτερον, όπως και εγώ γνωρίζετε εξίσου καλά ότι για τους κοινικούς είναι η, μια προσπάθεια να επανέλθει η ισχύ η, συνθήκη ABM από την πίσω πόρτα. Ξέρετε ότι αυτή είχε υπογραφεί κατά περίεργο τρόπο από δύο κράτη. Το θέμα είναι μπορεί να επανέλθει η συνθήκη ABM από την πίσω πόρτα. Και δεύτερον, γνωρίζω τις δυσκολίες τουλάχιστον ένας από τους 28 συμμάχους θα έλεγε όχι. Και επίσης εμείς ως ΝΑΤΟ δεν έχουμε ιστορικό στο να περνάμε νομικά κείμενα από τα κοινοβουλιά μας για ακύρωση. Δεν είναι κάτι στο οποίο το ΝΑΤΟ έχει καλές επιδόσεις μέχρι τώρα κατόπιν. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είχαμε προσεγγίσει τόσο πολύ να ξεπεράσουμε τις σκιές μας από τα τελευταία χρόνια. Με τη Λισαβόνα υπήρξε η όθηση, τώρα όμως δεν τη βλέπω πια. Ελπίζω να επανέλθει, αλλά ποτέ δεν είχαμε πλησιάσει τόσο κοντά. Το βασικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα έλεγα ότι η συζήτηση, όπως τη βλέπουμε στον τύπο, είναι ψεύδο συζήτηση πολύ συχνά είναι ψευδή συζήτηση να πούμε ότι η πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ υπονομεύει την αποτρεπτική δύναμη της Ρωσίας, στρατηγική δύναμη της Ρωσίας. Και εσείς είπατε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ΝΑΤΟ. Αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από την πυραυλική άμυνα. Υπάρχει έλεγχος του διαστήματος στην υπόθεση αυτή, το παγκόσμιο χτύπημα, το Global Strike Όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό, αν τα δείτε, τότε αντιλαμβάνομαι την άποψη της Ρωσίας. Όχι αν δούμε μόνο την ε, πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι ένα ελάχιστο κομμάτι σε σχέση με την δυνατότητα υπονόμευσης της στρατηγικής αποτρεπτικής δύναμης της Ρωσίας. Τώρα, το επόμενο θέμα. Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα που τώρα αντιμετωπίζουμε είναι το αδιέξοδο στα έγγραφα στα οποία, επί των οποίων διαπραγματευόμαστε. Η κοινή ανάλυση, δεν ξέρω πόσες αναθεωρήσεις έχουν γίνει, νομίζω πάνω από 20. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο είναι γεμάτο κείμενο σε ε, διαγραφές, επισημάνσεις, και δεν είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές επειδή σε αυτές τις προτάσεις αντικατοπτρίζεται η διαφωνία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όπως βλέπουμε, έτσι βλέπουμε την έλλειψη πρόοδου και το γεγονός ότι τώρα είμαστε σταματημένοι. Και βεβαίως υπάρχει μια έκθεση της ολοκλήρωσης της άσκησης αυτή συντάχθηκε πέρσι και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για τον ίδιο λόγο. Η Ρωσία δίνει μία ερμηνεία ότι η άσκηση έγινε και το ακούσαμε και από τον αξιότιμο συνάδελφο ότι η άσκηση δείχνει ότι από κοινού είναι καλύτερα. Ενώ άλλοι από τους συμμετέχοντες λένε ότι είναι πάρα πολύ πρόημο αυτό το συμπέρασμα με βάση μία μόνο άσκηση. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω ασκήσεις για να διερευνηθεί το σύντημα. Με δύο λόγια αυτή είναι η κατάσταση στο σημείο αυτό. Τώρα όσον αφορά την απειλή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω για το Ιράν. Απλώς να πω ότι το ΝΑΤΟ δεν επισημαίνει, καταδεικνύει συλλογικά οποιαδήποτε χώρα, αυτό πρέπει να το πούμε. Η κυρία Κοπά νομίζω είπε ότι, ότι δεν μιλάμε για καρτούν, δεν μιλάμε για τον και Τζέρι, κάποιος κρύβει κάτι, κάποιος δείχνει κάτι άλλο κτλ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόοδο στον τομέα του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα όχι μόνο για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και επίσης υπάρχουν δηλώσεις αρχηγών κρατών που λένε ότι εάν αλλάξει η απειλή θα προσαρμοστεί και το ΝΑΤΟ και θα το μελετήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο αγνοήσαμε τελείως. Εν πάση περιπτώσει δεν κάνω καμία άμεση σχέση ε, σύνδεση με το Ιράν γιατί δεν υπάρχει ε, από το ΝΑΤΟ ε, συλλογική επισήμανση του Ιράν. Η προσέγγιση μας είναι ότι η πυραυλική άμυνα σημαίνει ότι θα μειωθεί, ότι δεν θα αυξηθεί ο κίνδυνος από πυραυλικές επιθέσεις. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση για το άρθρο 5 για την έρευνα, για την ε, διοίκηση και τον έλεγχο. Για μένα είναι μια τεχνητή ψευδής συζήτηση. Καμιά φορά ακούω τους συμμάχους να λένε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με τη Ρωσία γιατί δεν είστε μέλος του ΝΑΤΟ. Το παραδέχομαι. Η Ρωσία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το επιχείρημα εγώ. Όμως πρέπει ταυτόχρονα να επισημάνω ότι και η Ρωσία πολύ συχνά λέει το ίδιο πράγμα. Ότι πολύ συχνά έχουμε ακούσει δηλώσεις υψηλόβαθμων Ρώσων που λένε ότι κανένας άλλος εκτός από τη Ρωσία δεν είναι υπεύθυνο για την άμυνα των ρωσικών εδαφών. Άρα και οι δύο πλευρές κάνουν τέτοιε δηλώσεις. Λένε οι μεν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λόγω του άρθρου 5 και η Ρωσία λέει ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά μας. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα βασικά ζητήματα εξακολουθούν να είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει. Και επανερχόμαστε σε αυτά που ακούσαμε, σε αυτά που είπαμε, να ξεπεράσουμε τη σκιά μας ο καθένας, τους φόβους μας που δεν το έχουμε πετύχει. Και θα κλείσω με ένα θέμα τα βασι... οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε Νικολάη είναι η, το αδι, ο αδιέρετος χαρακτήρας της ασφάλειας και η, ίση βάση. Ε, έχω ακούσει τους όρους αυτούς επανειλημμένως από Ρώσους αξιωματούχους τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι τα οποία είναι η σημεία αυτά τα οποία πρέπει να τα επισημάνουμε. Και όχι μόνο μέσω της πυραυλικής άμυνας πρέπει και αλλιώ να τα χειριστούμε, να, τα, να ασχοληθούμε μαζί τους. Γιατί το θέμα δεν είναι τόσο πολύ τώρα να βρούμε συμφωνία για την πυραυλική άμυνα, αλλά να βρούμε μια συμφωνία εμπιστοσύνης και να, ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και τώρα λοιπόν θα δώσουμε τον κύριο Φρανς Κλέχεκ για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι βεβαίως ε, είναι δύσκολο να ολοκληρώσει κανείς ε, και να παρουσιάσει όλα αυτά που ελέγχθησαν, τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν. Αλλά εγώ εντόπισα τουλάχιστον τρία στοιχεία και θα ήθελα να προσθέσω και κάποιες δικές μου απόψεις. Όπως ε, υπογράμμισαν αρκετοί, η συνεργασία οι δραστηριότητες που αφορούν στη συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια οδηγήθηκαν σε διέξοδο. Μετά την ε, ανταλλαγή δηλώσεων, ε, την πρώτη επιχείρηση, ε, την κοινή γλώσσα, τίποτα πλέον δεν προχώρησε και ακούγοντας και τους δύο μιλητές δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα ε, τα επόμενα έτη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η εμπιστοσύνη κάποια στιγμή σταματάει να υπάρχει. Άρα δηλαδή κάτι υπάρχει πίσω από αυτό, πολύ σημαντικότερο, πολύ μεγαλύτερο, που εμποδίζει να επεκταθούν δραστηριότητες. Κυρία είπε ότι θα, ήταν, θα είχε ενδιαφέρον να το εξετάσουμε αυτό περισσότερο διεξοδικά. Αναφέρθηκε επανειλημμένα το δυναμικό περιβάλλον ασφάλειας. Υπάρχει απειλή. Θα υπάρξει αύριο, μήπως μετά από 10 χρόνια σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί, να ισχυριστεί κανεί κάτι τέτοιο. Θέλω όμω να σα υπενθυμίσω ότι η πυραυλική άμυνα δεν είναι εύκολη και σε επίπεδο τεχνολογία. Υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία, ε, κυρίω ε, όσον αφορά του πυράβλου μεγάλου βεληνικού. Ε, σε αυτή την περίπτωση, τη συμφωνία με το Ιράν ε, για, για τον πυρονικό αφοπλισμό ή τον έλεγχο των πυρηνικών. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να ανασταλεί το ε, πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας και πρέπει να γνωρίζουμε τι θα συμβεί τους αμέσους επόμενους ε, μήνες, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας του Ιράν. Η ανάπτυξη αναπτικής, ε, αμυντικής δυνατότητας και επιθετικής ε, δυνατότητας αυτά χρειάζονται χρόνο, δεν γίνονται μέσα σε λίγους μήνες ή το πολύ ένα χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, πριν παρατηθούμε από κάτι, να έχουμε κατά νου, να παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η ε, ανάπτυξη λοιπόν αφορά και τις δύο πλευρές και το να σταματάει κανείς ένα πρόγραμμα ε, απλά και μόνο επειδή εμφανίζεται κάποιο πουλί στον ουρανό, μα δεν σημαίνει αυτό ότι επίκειται η άνοιξη. Ας δούμε λιγάκι τους ε, τομείς όπου μπορεί να υπάρξει οικοδόμηση εμπιστοσύνης πέρα δηλαδή από στενά το πλαίσιο της πυραυλικής άμυνας. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω να προτείνω. Εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει στην ε, στρατιωτική συνεργασία για αστικούς ε, σκοπούς. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η δυνατότητα κατάρριψης ε, πυράβλων προφανώς και έχει συνέπειες στο έδαφος. Δεν είναι ο στρατός που θα ξεκαθαρίσει εκ των την κατάσταση, αλλά η πρώτη που θα πρέπει να ε, ανταποκριθούν, να λάβουν τα μέτρα τους, ε, είναι η ε, πολιτική προστασία. Εδώ λοιπόν το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι εταίροι θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανταλλάξουν απόψεις, να οργανώσουν επιχειρήσεις, να οργανώσουν το σύστημα ελέγχου και άμυνας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούν να γερθούν μεταξύ αυτών και τα πυρηνικά. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπως έτσι ε, λέχθησαν αυτά σήμερα και προσέτσα βέβαια και εγώ κάποιες δικές μου απόψεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις που κάνατε. Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι είμαι σίγουρος ότι το, μέλλον αυτό το θέμα αυτό θα ξανασυζητηθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα μετά από αυτές τις ε, πληροφορίες που αντιλάγησαν και τώρα νομίζω ότι έχουμε μάθει βέβαια περισσότερα για τα συστήματα. Πάμε στο επόμενο θέμα και αυτό βρίσκεται από τον ίδιο χώρο ένα αντιπυραυλικό σύστημα για την Ευρώπη, ο πολιτικός και ο στρατηγικός αντίκτυπός του. Έκθεση του κυρίου Σάμπο Τέρχο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mm. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα κάνω τις ε, παρατηρήσεις μου στα φινλανδικά, οπότε αν θέλετε φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Niin, Σας ευχαριστώ. Στην έκθεση αυτή προσπαθώ να κάνω μια να δώσω μια εικόνα του αντιπυραυλικού συστήματος της Ευρώπης, τις δυνατότητες, τις απειλές και προσπαθώ να διατηρήσω μια ουδέτερη στάση. Η πραγματικότητα μιας πυρηνικής απειλής είναι πάντοτε παρούσα στην Ευρώπη ακόμα και αν έχει μειωθεί. Ακόμα και αν είναι ελάχιστη μια τέτοια απειλή, θα πρέπει πολύ σοβαρά να την αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, ακόμα και αν τα ευρωπαϊκά αντιπυραυλικά συστήματα μπορεί να προκαλέσουν τα πολιτικά πάθη, ελπίζω πως θα μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα αυτό από τεχνική και ρεαλιστική άποψη. Τι σημαίνει αυτό, ότι για να υπάρξει ένα σύστημα λήψης αποφάσεων, αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ε, ερευνητικά στοιχεία, σε αναλύσεις που έχουν ε, ε, γίνει σε σχέση με το κόστος και το όφελος ενός τέτοιου συστήματος. Αν λάβουμε την απόφαση να οικοδομήσουμε ένα αντιπυραυλικό σύστημα, ποτέ δεν, πρόκειται, πρέπει να πρόκειται μάλλον για μια ιδεολογική οικοδομή, ένα οικοδόμημα τέτοιου τύπου. Θα πρέπει βασικά να ασχοληθούμε μόνο με το θέμα κόστους οφέλους, γιατί πρόκειται για ένα σχέδιο πολύ πολύ δαπανηρό και πιστεύουμε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε αρκετά ερευνητικά στοιχεία ουδέτερα ώστε να βασιστούμε σε αυτά και να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στην έκθεση αυτή μια πιο ε, λεπτομερή διευκρίνηση επί τη βάση της οποίας να μπορέσουμε να λάβουμε πιο ρεαλιστικές ε, αποφάσεις ε, προσπάθησα να κάνω ένα πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε με βάση τις υπάρχουσες αναλύσεις, πώς θα κατασκευαστεί, ποιες είναι, ποιες είναι ο στρατηγικός αντίκτυπος, ποιος είναι η επίπτωσή του στην φύση της κοινή άμυνας στην Ευρώπη και ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις απέναντι στην κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος. Ακούσαμε κάποιες ε, προηγούμενες αντιδράσεις ήδη κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Ε, η συνεργασία με τη Ρωσία θα ήταν πολύ κρίσιμη για να σταθεροποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα και οι επιπτώσεις του. Επίσης εξαιρετικά σημαντικό θα ήταν να θυμηθούμε πως αν δεν υπάρχει ένα σύστημα, μάλλον μια ε, αλυσίδα αποτελεσματική για τη λήψη αποφάσεων μια σωστή αλυσίδα διοίκηση, θα υπάρξουν προβλήματα. Αυτά έχω να σας πω ε, και περιμένω τις αντιδράσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Thank ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κοιτάξτε, τώρα βρίσκομαι σε μια περίεργη κατάσταση, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι και σκιώδη ηγητή αυτή τη έκθεση ε, για το ΕΛΚ. Και εγώ θα μιλήσω πολωνικά, γιατί υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί όροι και προτιμώ να μιλήσω στα πολωνικά. Αν έχετε καλοσύνη να βάλετε ακουστικά σας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Τάρκο. Ε, πιστεύω ότι η δομή της έκθεσης είναι καλή. Η έκθεση έχει συνταχθεί με έναν ιδιαίτερα περιεκτικό, ουσιαστικό τρόπο, αλλά θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες και ελπίζω να συμφωνήσετε με την τελική μορφή που θα λάβει η έκθεση. Η επικεφαλίδα είναι αντιπυραυλική ασπίδα για την Ευρώπη, πολιτικές ε, και στρατηγικές ε, προεκτάσεις. Έχοντας όμως κατά νου την κατάσταση που επικρατεί, η αντιπυραυλική αυτή ασπίδα με βάση ε, τις αμερικανικές προδιαγραφές, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση. Ε, έχω αναλύσει το σχέδιο της έκθεσης και έχω εξάγει αρκετά συμπεράσματα. Πρώτον, ως σκιώδης συγητής πιστεύω ότι διαβάζοντας κανείς την έκθεση μπορεί να αποκομίσει την εντύπωση ότι περιγράφει μια κατάσταση όπου η Ευρώπη οικοδομεί τη δική της αντιπυραυλική ασπίδα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Λισαβόνα και το Σικάγο δηλαδή να υπάρχει προστασία για το σύνολο της Ευρώπης ε, γιατί τώρα ε, το σύστημα βασίζεται στην, ε, στις αμερικανικές ικανότητες. Η εθνική ικανότητα θα χρησιμοποιείται και θα ενταχθεί στο κοινό σύστημα ελέγχου. Το σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται, θα είναι λειτουργικό. Αυτή είναι η πρώτη δήλωση που έγινε στο Σικάγο Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επισημαίνουμε την διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η αντιπραυλική ασπίδα είναι μια αμυντική ικανότητα η οποία συμβαδίζει με την επιθετική ικανότητα. 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Σικάγο αποφάσισαν το σύστημα αυτό να μπορεί να προστατεύσει την επικράτεια του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που είναι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, της ε, υπηρετικής Ευρώπης, ε, η Γρυλανδία, η Τουρκία και τα νησιά της Μάνχης. Υπάρχει και το εδάφιο Β που είναι ένα σύμβολο συμμετοχής ε, των Ηνωμένων Πολιτειών στην άμυνα της Ευρώπης. Ε, εδώ θα πρέπει να το αλλάξουμε και να πούμε συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ε, σε θέματα του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν και εδώ παραθέτω, δεν μπορούμε να λέμε ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για να προστατεύσει μια συγκεκριμένη χώρα, κυρίως αυτήν στην οποία είναι εγκατεστημένο. Το σύστημα αυτό θα προστατεύει χώρες ε, όπως την Πολωνία και τη Ρουμανία και βεβαίως ε, οι ίδιες αυτές εγκαταστάσεις μπορούν να προστατεύσουν και οι γειτονικέ χώρες. Στο άρθρο υπαριθμών 2 ο εισηγητής λέει ότι με βάση αποφάσεις που ελήφθησαν από τους Αμερικανούς αυτό το οικοδόμημα του ΝΑΤΟ δεν θα αφορά ε, τα συστήματα αναχέτησης ε, της Ευρώπης όπου αυτά τα συστήματα υποτίθεται θα αναχαιτίζουν ε, πυράβλου πρώτη γενιά όπω αυτοί που εκτοξεύονται παρήματο χάρη από τη Μέση Ανατολή. Άρα ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα προστασίας τουλάχιστον σε αμερικανικό έδαφος. Επίσης αναφέρεται ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα, η πέμπτη φάση και άρθρο 15. Αυτή η σύσταση μπορεί να ισχύει μόνο σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι πρέπει να φτιάξει μια αντιπυραυλική ασπίδα για απειλές όπως αυτές που μπορούν να προέρχονται ενδεχομένως από τη Βόρεια Κορέα. Εμείς καταγγέλουμε ε, τις ε, προσπάθηση της ε, Βόρειας Κορέας να εμφανίσει ένα νέο όπλο αλλά μοιάζουν και η εμβέλειά του να είναι περιορισμένη. Όσον αφορά την απειλή από το Ιράν δεν μιλάμε για διπηρετικούς πυράβλους αλλά μιλάμε για πυράβλους μέσου βεληνικούς διότι η χώρα αυτή ε, αν μας επιτεθεί ε, με πυράβλους μέσου ελληνικούς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους και η τρίτη φάση της αντιπυραυλικής ασπίδας ε, θα η τρίτη αυτή φάση ε, δεν θα ισχύει για βαλιστικούς πυράβλους πρώτης γενιάς διατύπωση, κάτι που συζητήσαμε πρόσφατα ε, σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ αμυντικά. Ε, παρότι βέβαια αυτή η ασπίδα δεν αφορά ιδιαίτερα τη Ρωσία, πιστεύω ότι το να καλέσουμε τη Ρωσία να συμμετέχει στην οικοδόμηση αυτού του συστήματος, άρθρο υπαριθμών 7, νομίζω ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάτι τέτοιο είναι πολύ πρόωρο. Το ΝΑΤΟ θέλει συνεργαστεί με τη Ρωσία, αλλά μιλάμε για δύο ε, διαφορετικά συστήματα, ανεξάρτητα. Το ένα ανήκει στο ΝΑΤΟ, το άλλο στη Ρωσία. Στο Σικάγο προσφέραμε στους Ρώσους ε, τη διαφάνεια, αλλά η διαφάνεια είναι και πρέπει να είναι αμφίδρομη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ενθαρρύνουμε τους Ρώσους να προτιμάσουν επικοδομητική προσέγγιση δεν υπάρχει καμία απειλή για το ε, αποτρεπτικό σύστημα του ΝΑΤΟ. Κατά την άποψή μου εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα άρθρο μετά τις ε, συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γενέβη διότι οι πυραυλικές ασπίδες ε, οικοδομούνται ή υπήρξαν κυρίως για την απειλή από το Ιράν και με βάση τη νέα όμως συμφωνία μπορούν να εμπλουτίσουν το ουράνιο μέχρι 5% και ότι είναι πάνω από το 5% εμπλουτισμένο με ουράνιο πρέπει να καταστρέφεται πριν επιβάλλουμε εμείς κυρώσεις. Και νομίζω η τελευταία παρατήρηση είναι η εξή. Είναι πολύ σημαντικό ε, να ε, υπάρχει σωστή κατανομή της νομολογίας και των ικανοτήτων αν δεν υπάρχει άμεση απειλή από τρίτη χώρα η ε, βοήθεια πρέπει να προσφέρεται κυρίως από το ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 5 της ε, Συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Η κυρία Κοπά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ισκιώδης εισηγητής μας ε, είναι σήμερα μιλητής αλλού και γι' αυτό θα σας μεταφέρω κάποια μηνύματά του, τη μηνύματα της ομάδας. Καταρχήν είδαμε το σχέδιο έκθεσης του κ. Σαμποτέρο ως έγγραφο εργασία με και ως ε, σημείο αφετηρίας για συζήτηση στην Υποεπιτροπή. Θεωρούμε ότι το κείμενο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και να αλλάξει σημαντικά για τρεις τουλάχιστον λόγους το κείμενο αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρώτον, η παρούσα πρόταση μοιάζει ότι δεν είναι σωστή ως προς τα περιστατικά. Ο κ. Σταρό θεωρεί ότι η αμυντική άμυνα του ΝΑΤΟ θα προσφέρει προστασία για βασικά στοιχεία του, ε, ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα καλύπτει όλοι τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Αυτό αναπτύχθηκε, αλλά Όλα αυτά έχουν προκαλέσει υποστήριξη για μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα. Η υποστήριξη για μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα είναι αυτή τη στιγμή όνειρο ε, δεδομένων των περικοπών και της οικονομικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Επίσης, δεν γνωρίζουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, η ομάδα, σας, ε, ε, η ομάδα μας επανειλημμένος και διαρκώς στηρίζει όλες τις πρόσφατες αναφορές και τις εκθέσεις από τη CSTP και τη CFCP και επίσης την σημασία της διατλαντικής σχέσης. Αυτά δεν καλύπτονται στο το σχέδιο έκθεσης που καλύπτει με το βασικό στοιχείο της άμυνας, την πυραυλική άμυνα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ε, να υποβάλουμε αλλαγή που θα τονίζει την συμπληρωματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το θέμα της συνεργασίας με τη Ρωσία για την πυραυλική άμυνα. Είναι γνωστό ότι η σχέση είναι πολύ σύνθετη και όχι όπως παρουσιάζεται στην πρόταση αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρέπει να, να χρησιμοποιηθεί ο όρος βαλιστικής πυραυλικής άμυνας. Η ασπίδα είναι ένας όρος που προκαλεί σύγχυση. Επίσης, υπάρχει μια διατύπωση που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Στην παράγραφο 4 ας πούμε παραθέτω παράγοντες που δεν ε, εμπίπτουν, που δεν τηρούν ε, την παραδοσιακή αντίληψη του ορθολογισμού. Δεύτερο σημείο της παραγράφου 7. Παραθέτω για ε, χιλιάδες άνεργοι πυρηνικοί επιστήμονες πρώην Σοβιετική Ένωση αποτελούν διαρκή απειλή για τη μεταφορά επικίνδυνων πληροφοριών. Αυτό είναι ανεπαρκής διατύπωση ενό τέτοιου κειμένου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το ε, τροποποιήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πάσκο ε, είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον εισηγητή, τους άλλους σκιώδης και τη γραμματεία για να ξαναρχίσει η συνεργασία για μια έκθεση που ασχολείται με ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόπα. Κύριε Κρόνμπεκ, παρακαλώ. Thank you. First of all, I agree with the rapporteur, Sam Poterho, that, that uh, the analysis of the... Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει η ανάλυση να βασιστεί μάλλον η μελέτη της αντιπυραυλική άμυνας θα πρέπει να βασιστεί σε αναλύσεις. Το θέμα είναι τι ανάλυση χρειαζόμαστε. Νομίζω πως η κύρια ιδέα της Ένωσης όσον αφορά την άμυνα είναι η Ρούσεων. Και στην ουσία η πυραυλική άμυνα δημιουργεί, προκαλεί συγκρούσει σε τοπικό επίπεδο από τα ραντάρ είναι τα πρώτα τα οποία στοχεύονται και δημιουργεί, προκαλεί σύγκρουση σε διεθνές επίπεδο και το βλέπουμε αυτό ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Εγώ θα ήθελα να δούμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πυραυλική άμυνα και την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και των πυραυλικών τεχνολογιών. Είναι βέβαιο πως η πυραυλική άμυνα είναι ένα εργαλείο για την μη εξάπλωση, έτσι λέγεται, αλλά είναι λάθος. Μπορούμε να δούμε τι Κίνα, γιατί ο ειρηνικός καλύπτεται από πυραυλική άμυνα, ενώ το κινέζικο πυρηνικό ε, οπλοστάσιο όχι ε, περιορίζεται, έτσι, αλλά επεκτείνεται. Μπορούμε επίσης να το δούμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος της, ε, της δημιουργίας μάλλον πυραυλικής άμυνας στη Μέση Ανατολή και άρα και η εξάπλωση της ε, πυρηνικής ενέργειας αλλά και των πυραυλικών τεχνολογιών. Γι' αυτό νομίζω πως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η μη εξάπλωση είναι ένα θέμα χωριστό από την πυραυλική άμυνα. Έπειτα, το θέμα των απειλών. Το Ιράν έχει αναφερθεί ως απειλή, αλλά αυτό ανεφέρθηκε στην στο αρχικό και στα αρχικά κείμενα του ΝΑΤΟ, αφαιρέθηκε γιατί η Τουρκία αποφάσισε πως το Ιράν δεν ήταν απειλή και νομίζω πως η επίσημη εικόνα των απειλών του ΝΑΤΟ είναι 30 χώρες που μπορούν να στείλουν ε, πύραυλους στην Ευρώπη. Άρα έχουμε να κάνουμε με πιο περίπλοκη απειλή και όχι, με ένα απλό, και όχι μόνο με το Ιράν. Αν και ελπίζω ότι θα πάψει να υφίσταται και η απειλή του Ιράν. Στην έκθεση γίνεται μια πρόταση για την εξέβρεση θεσμικών ρυθμίσεων με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συνεργαστούν οι τρεις αυτοί. Η συζήτησή μας εδώ λοιπόν γίνεται πριν αυτή η έκθεση να επικυρώσει ότι σήμερα δεν υφίσταται οι προϋποθέσεις που θα προωθούσαν ε, την ιδέα μιας ε, διαθεσμικής συνεργασίας. Μάλιστα, η διαθεσμική συνεργασία για την οποία υπήρχαν οι προϋποθέσεις πριν από δύο χρόνια, πλέον δεν υπάρχει. Και υπάρχουν λόγοι για, γι' αυτό και παρουσιάστηκαν εδώ. Η έκθεση εξετάζει τους παράλογους ε, παράγοντες, εκείνους τους ηγέτες που δεν έχουν να χάσουν τίποτα και μπορεί να αρχίσουν να στέλνουν πυρηνικά ή πυράβλους στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω πως αυτό είναι πολύ δαπανηρό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους παράλογους παράγοντες. Δεν θεωρώ πως η πυραυλική άμυνα είναι η λύση για την αντιμετώπιση των τρελών δικτατόρων. Το κόστος της πυραυλικής άμυνας βέβαια είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του Σαν Ποτέρχο για μια ανάλυση κόστος ωφέλειας. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο επί ουδέτερης βάσης, αλλά θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Και επίσης θέμα είναι και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν σκεφτεί ότι η θα σταθεί σε, αυτά, σε αυτή την κατάσταση ενώ οι ΗΠΑ αποσύρονται από την Ευρώπη δεν είναι ρεαλιστικό να σκεφτεί κανεί ότι οι Αμερικανοί θα καλύψουν κάποιο κομμάτι του κόστου, οποιοδήποτε κομμάτι του κόστου. Τώρα, αφού οι χώρε οι Ευρωπαϊκέ χρησιμοποιούν τι αμυντικέ του δαπάνε και τι περιορίζουν και μιλάμε για συγκέντρωση και κατανομή, pooling and sharing, θα ήταν λογικό ε, να μιλήσουμε για να επενδύσει σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει ακόμα και σωστά λέει η έκθεση ότι πρέπει να μελετηθεί και η τεχνολογική σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος. Δεν είναι βέβαιη ούτε αυτή. Και έπειτα υπάρχει και κάτι στην έκθεση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γινόταν μια πραγματική ένωση αμυντική εάν φτιάχναμε την αντιπυραυλική ένωση. Νομίζω όπως η τεχνολογία και η πολεμική τεχνολογία ποτέ δεν έχει οικοδομήσει ενώσεις, μόνο πολιτικές, η πολιτική ένωση μπορεί να σταθεί. Ευχαριστώ η κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια ε, σε αυτή την έκθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντική και δεν μπορώ και εγώ να μην πω τίποτα. Διάβασα λοιπόν την έκθεση ε, και θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε πριν από κάποια χρόνια όταν ε, η όλη αυτή η ιδέα του να εγκατασταθούν συστήματα ραντάρ αντιπυραυλικά στην Ευρώπη τότε είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο κατά πόσο να έπρεπε να το δεχθούμε αυτό το πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα συνδεόταν ή όχι με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος και τα θυμάμαι αυτά αρκετά καλά και γνωρίζω εξίσου καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Φοβάμαι λοιπόν ότι παρά τις ε, καλές ε, προσπάθειες η έκθεση τελικά δεν αναφέρει με ακρίβεια το πόσο περίπλοκο είναι το όλο θέμα. Το υποτιμά κατά κάποιον τρόπο. Επίσης Νομίζω στο σημείο υπερθμών 12 της έκθεσης εκεί αναφέρεται ότι αν τελικά αποδειχθεί ότι το σύστημα είναι αποτελεσματικό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει αυτό το σύστημα. Και δεν ξέρω αν συμφωνούμε όλοι μας να αναφέρεται αυτή η άποψη τόσο ξεκάθαρα. Και μια άλλη παρατήρηση θέλω να κάνω. Φοβάμαι ότι ο συνάδελφός μας είναι υπεραισιόδοξος, κυρίως εκεί όπου αναφέρει ότι είναι πολύ εύκολο το να υπάρξει ένα αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι χώρες εκτός του ΝΑΣΟ, ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θα μπορούσαν να συνεργαστούν για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Εγώ λοιπόν σας ε, λέω ήδη τώρα ότι θα καταθέσουμε μία σειρά τροπολογιών. Ε, θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τη δική μας θέση, γενικότερα το όλο θέμα. Με πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση πρέπει να σας πω ότι η δική μας ε, η πολιτική ομάδα έχει έντονες επιφυλάξεις για όλα αυτά που αναφέρονται στην έκθεση. Ο κύριος ε, Τάνοκ. Κοιτάξτε, ε, εγώ δεν, ούτε κι εγώ είμαι σκιώδης ηγητής ε, της ομάδας μου. Είμαι συμπληρωματικό μέλος αυτής της επιτροπής, αλλά νομίζω ότι η δική μου η ομάδα στηρίζει αυτή την έκθεση. Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ της τεχνολογίας της αντιπυραυλικής ασπίδας για να αποτρέψουμε ένα κακοποιό κράτος ή οποιονδήποτε δεν θέλω να αναφέρω, να ονοματίσω, αλλά θέλουμε να εμποδίσουμε οποιονδήποτε να επιτεθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ότι αυτό μπορεί να το κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου είναι σενάριο φαντασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διμερές επίπεδο και με το ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με θέματα κοινή ασφάλειας ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος. Αυτά που γίνονται στο Μαλί ε, με την πειρατεία, όλα αυτά καθιστούν ακόμα πιο σημαντική την ε, στρατηγική αντιπυραυλική άμυνα. Ε, θα στηρίξουμε την έκθεση, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη παράγραφος που με ενοχλεί. Εκεί όπου αναφέρεται ότι το Πακιστάν ε, θεωρείται ότι απειλείται από τη Βόρεια Κορέα και θυμάμαι ότι γύρω στο 2000, το 99, όπου ήταν το εξελέγει, τότε υπήρχε μια πολύ περίεργη ιστορία με τα όπλα στο Πακιστάν και ο πρέσβης ο Πακιστανός τίμωσε πάρα πολύ μαζί μου γιατί εγώ τα καταγγείλα, ε, αυτά δημοσιεύτηκαν. Εντάξει, εγώ ζήτησα συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσίασα. Εν τόσο, όλα αυτά τώρα είναι παρελθόν και ξέρουμε ότι το Πακιστάν ε, έχει την ε, πυρηνική όπλα. Ο ίδιος συνελήφθη πριν από κάποια χρόνια. Το Πακιστάν ισχυρίζεται το αντίθετο. Δεν ξέρω όμως αν μεταξύ υπάρχουν νέα στοιχεία. Γιατί υπάρχουν πολύ ε, σοβαροί πενιγμοί και θα ήθελα να ξέρω τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε να συντάξετε την παράγραφο 7 της έκθεσης. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Μισό λεπτό, αν έχετε καλοσύνη να είστε και σύντομο, γιατί είμαστε λιγάκι καθυστερημένοι στην ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, η ομάδα μα είναι αντίθετη ε, με την έκθεση, γιατί γενικά είμαστε αντίθετοι με αυτό το σύστημα. Θεωρούμε ότι δεν προσφέρει τίποτα. Αντιθέτω, αυξάνει την ανασφάλεια και τον ανταγωνισμό για του εξοπλισμού. Χώρια που Βέβαια η έκθεση προσπαθεί να μειώσει λίγο τις επιπτώσεις μελλοντικά. Μιλάει για ένα μικρότερο σύστημα τώρα και στο μέλλον θα δούμε τι θα γίνει, αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι θα ακολουθήσει. Τέλος, νομίζω ακριβώς αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ε, η συμφωνία δηλαδή με το Ιράν όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα είναι ο δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων και αν έχουμε τέτοιου είδους ανησυχίες θα έπρεπε να υπάρχει ένας γενικός πυρηνικό αφοπλισμός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Κύριε Τέρχο, θέλετε να απαντήσετε, να σχολιάσετε ε, όλα αυτά που ακούστηκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ακριβώς αυτό προέβλεπα. Όλοι έχουν ε, μια ισχυρή άποψη για το πώς θα πρέπει να, είναι το, να τεθεί το ζήτημα θεωρούσα ότι δεν έχω εγώ ε, ξεκάθαρη ε, ισχυρή άποψη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό το έγγραφο στο μέλλον. Όλα, αυτά μπορώ να πω μόνο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά μετέπειτα. Όταν ήδη θα έχουν υποβληθεί και κάποιες τροπολογίες για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θέλει να προχωρήσει την έκθεση κάθε πολιτική ομάδα. Όπως σας είπα, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε λογική πρόταση, ήδη το είπα αυτό κατά την εισαγωγική μου ομιλία και άρα εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο ότι τελικά η έκθεση θα είναι καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των σκιωδών εισηγητών μπορώ να δηλώσω ότι θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Τόργο. Και θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 7η Ιανουαρίου, Τρίτη, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στις 12 το μεσημέρι. Είναι λοιπόν εργασί... Ε, διακοπές εργασίας στο σκι μαζί με... θα πάτε για σκι μαζί με την έκθεση. Μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση σήμερα. Έχουμε ακόμα ένα ε, ενδιαφέρον ζήτημα. Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας και μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε δύο μιλητές, τον κύριο Walter Stevens, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και τον ε, αντιστράτηγο Wolfgang Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να είχα μάθει το όνομά σας προηγουμένως, λέει ο Πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε κύριοι, το σύστημα αυτό συζητείται εδώ και μήνες, δύο μήνες, αλλά προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο την ε, διάσκεψη κορφής του Δεκεμβρίου. Είναι λοιπόν ε, πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα και τι να περιμένουμε τελικά. Λοιπόν, ο κύριος Στίβενς, καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συναντηθώ με την Επιτροπή. Έχω ήδη συναντηθεί στο παρελθόν επανειλημμένος όταν ήμουν διευθυντής της CMPD και τώρα ως πρώτη φορά ως πρόεδρος της PSE. Ε, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα. Όλοι θεωρούμε πολύ σημαντικές τις επαφές μας με το Κοινοβούλιο και τις πολύ σημαντικές εκθέσεις που κάποια μέλη της Επιτροπής έχουν υποβάλει κυρίως στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας και ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας είναι πολύ καλές εκθέσεις. Όπως είπα, η PSC ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και με την CSTP. Σήμερα λοιπόν θα πω δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας, το οποίο είναι ε, σε προετοιμασία, καταρχήν για την προετοιμασία και την ουσία και κατόπιν θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που αφορούν στις ε, αποστολές της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της CSDP. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι βάζοντας το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ο Herman Van Rompuy έχει δημιουργήσει μια τρομερή ένα τρομερό αντίκτυπο. Το 2013 ήταν μια χρονιά του CSDP, της, CSDP, της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας συνεισφορά με τις ε, εξαιρετικές εκθέσεις του κ. Μπρόκ και τις άλλες. Όλα αυτά είχαμε την ενδιάμεση έκθεση που μπόρεσε να σχολιάσει ο υπουργό στο Βίλνιους και αργότερα την επίσημη έκθεση που οδήγησε την τελική έκθεση της καθιάστων η οποία ήταν εξαιρετικά ευπρόσδεκτη από τους υπουργούς ως εξαιρετική βάση συμπερασμάτων. Τώρα πλέον τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν με κάποια δυσκολία, τελική ευθεία και είναι ουσιαστικά. Κάποιοι λένε ότι είναι κάπως μακροσκελή, 17 σελίδες, 30 ή 40 παράγραφοι που αφορούν τις τρεις ομάδες. Την αποτελεσματικότητα και την ε, εμφάνιση των δυνατοτήτων της κοινή ε, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Επίσης υπάρχουν όμως και προτάσεις που αφορούν τη βιομηχανική βάση της άμυνας. Και εδώ έχουμε αρκετά ουσιαστικά στοιχεία και επίσης έχουν σχέση και με την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφάλεια και την άμυνα που ε, δόθηκε στη δημοσιότητα ταυτόχρονα και είναι αξιο, σημείο το ότι στις τελευταίες εισηγήσεις και αυτό ήταν και το θέμα των Υπουργών, το θέμα αφορούσε τη βιομηχανία. Τα τρία προβλήματα ήταν το πεδίο της βιομηχανικής βάσης, για την άμυνα. Δεύτερον, είχε σχέση με το αν θα υπάρξει κάποια προστασία της αγοράς, ίσες ευκαιρίες, αν όλοι θα έχουν μερίδιο της πίτας και επίσης περισσότερος ανταγωνισμός ελεύθερη ανοιχτή αγορά. Και το τρίτο είχε σχέση με το ότι βεβαίως χρειαζόμαστε κίνητρα για συνεργασία στο τομέα, στον τομέα των δυνατοτήτων, αλλά άλλοι είπαν ότι πρέπει να δώσουμε και οικονομικά κίνητρα όπως είναι εξαίρεση από το ΦΠΑ κτλ. Αυτά είναι τα τρία-τέσσερα θέματα που θα εξακολουθήσουν να απασχολούν τους υπουργούς εστάλθηκαν στην Κορεπέρ και πάλι, αλλά γρήγορα βρέθηκε η λύση. Τώρα, μετά από όλα αυτά και αυτή την τα αρκετά εκτεταμένα και ουσιαστικά πράγματα, αρκετά φιλόδοξα, ίσως όχι τόσο όσο θα θέλατε εσείς, αλλά και αρκετά ρεαλιστικά. Έχουμε τα μακροσκελή συμπεράσματα όπου το γραφείο του Φαν Ρομπέι θα διατυπώσει συντομότερα και τα οποία θα προκινηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων κλπ. Θα παραμείνει πίεση ε, στην, μέσα στο σύστημα γιατί θα συναντηθούμε με το Van Rompuy σε λίγες μέρες. Αυτά τα συμπεράσματα είναι ουσιαστικό κείμενο. Σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση ανάμεσα στα τρία κομμάτια. Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις, βεβαίως, χρειαζόμαστε δυνατότητα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε και βιομηχανία να την αναπτύξει τη δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, σημαντικό είναι επίσης ότι δεν υπάρχει νέα στρατηγική, σαφώς. Αλλά υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο που περιγράφουν τα συμπεράσματα. Αναφέρονται σε νέες απειλές, ε, παλές, ε, απειλές το γεωστρατηγικό περιβάλλον, την έλλειψη χρηματοδότησης για τις δυνατότητες λόγω της ύπαρξης των οικονομικών προβλημάτων. Αυτό είναι το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο όλα συμβαίνουν. Τρίτον, υπάρχει σαφής δέσμευση πολιτική δέσμευση για την ασφάλεια της Ευρώπης και ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πάροχος ασφάλειας. Είναι σημαντικό που το διαπιστώνουν αυτό οι ηγέτες. Τέταρτον, εάν η Ευρώπη πρέπει να είναι πάροχος ασφάλειας, υπάρχει και ένα θεματολόγιο για το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Δεν είναι το πώς μόνο, αλλά όχι το τι, αλλά και το πώς θα το πετύχουμε αυτό μέσω δυνατοτήτων, μέσω της βιομηχανίας από το γεγονός ότι σημασία έχει η άμυνα, άρα πρέπει να υπάρχει αμυντική δυνατότητα και επίσης υπάρχουν θέματα ε, θαλάσσιας, υπάρχει η σχέση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, οι αρμοδιότητες, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Φυσικά όλες οι δυνατότητες, υπάρχουν τα ε, εμβληματικά σχέδια όπως η η παροχή καυσίμων ή το RPS. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι μια σοβαρή δέσμευση για βαθύτερη συνεργασία. Δηλαδή τα κράτη-μέλη και οι ηγέτες, τώρα υπουργοί, αλλά ελπίζουμε και οι ηγέτες, θα πούν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει βαθύτερη συνεργασία και αναγνώριση της αλληλεξάρτησης της ε, Τη άμυνα, ότι κανένα από μόνο του δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Χρειαζόμαστε όλοι μαζί. Και αυτό είναι μια σαφή δέσμευση που πρέπει να αναλυφθεί. Τώρα, πιο συγκεκριμένα. Αν δείτε, καταρχήν, υπάρχουν κάποια στρατηγικά στοιχεία, το στρατηγικό πλαίσιο. Αλλά στο πρώτο σκέλος, το CSDP, η βασική λέξη είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή πρέπει όλα να τα συγκεντρώσουμε. Και γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, συνεργάζονται για το κοινό ανακοινωθέν. Γίνονται βήματα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ας πούμε τις ε, αποστολές, πολιτικές αποστολές. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που πρέπει να ακολουθήσουμε, υπάρχουν όμως και οι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί που ε, έχουν παλιούς κανόνες οι οποίοι δεν είναι πάντα προσαρμοσμένοι στα νέα συστήματα. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Υπάρχει η, η, η ταχεία ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχουν οι, τα, οι Υπάρχουν τα battle groups τα οποία πρέπει να αυξηθεί ή, ε, να γίνουν πιο εμφανή, αλλά υπάρχει και η θαλάσσια στρατηγική, υπάρχει ο κυβερνοχώρος, υπάρχει η αλληλοσύνδεση της ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης, εσωτερικών υποθέσεων και εξωτερικών υποθέσεων. Υπάρχει το θέμα της τρομοκρατίας, θέματα μετανάστευσης, η νότια γειτονία, το θέμα των συνόρων, όλη αυτή η συνεργασία. Θα κάνουμε μία συνάντηση με τους συναδέλφους της Κόζη με δύο βασικά ζητήματα. Το θέμα των, της Συρίας, των ξένων μαχητών στη Συρία, γενικά, στη Συρία, ιδιαίτερα στη Συρία αλλά γενικά. Πάρα πολύ καλή υπήρχαν και οι υπουργοί εξωτερικών και το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε ήταν ακριβώς το θέμα της μετανάστευσης και των δυσκολιών στην νότια κοινωνία, ε, γειτονία, αυτά που γίνουν στη Λαμπετούσα κλπ. Όπως σας είπα, Έχουμε τον ανεφοδιασμό στον ε, αέρα, ε, ε, την ιδέα της διαρθωτικής συνεργασίας, πολύ σημαντικό κοινό σχεδιασμός, πάρα πολύ σημαντικός και δύσκολος. Η εντύπωση ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μοντέλα ε, τύπου ATTACK που συνδυάζουν ε, το σενάριες μεταφορές. Ε, αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα του πώς μπορούμε να δώσουμε κίντρα για αυτή τη συνεργασία με την ιδέα Μήπως θα μπορούσαν ας πούμε, αυτά τα προγράμματα συνεργασίας να περιορίσουν ε, τα, τις δαπάνες τους με συγκεκριμένες διευκολύνσεις ή ε, απαλλαγές από φορολογία και ούτω καθεξής. Τώρα και εδώ σε σχέση με την βιομηχανία και αυτό σχετίζεται γιατί αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η αγορά η αμυντική και εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Ναι ανταγωνιστική, ναι διαφανής, ναι πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό αλλά εγώ βλέπω ότι αυτοί που ανησυχούν περισσότερο για την προστασία δίνουν περισσότερη έμφαση στις μικρομεσαίες ε, ε, βιομηχανίες την ανάγκη γιατί αν θέλεις να αντιμετωπίσει αυτή την ε, καταγερματισμό, την ανάγκη για τυποποίηση και επιστοποίηση και εκεί βεβαίως χρειάζεται πρόοδος και τέλος πώς διατηρούμε την εμπειρογνωμοσύνη μας στην έρευνα και στην τεχνολογία. Να μην τη χάσουμε, γιατί έτσι μπορεί να προοδεύσει η βιομηχανία μας. Και τέλος, είναι κάπως δύσκολη συζήτηση ανάμεσα στην πολιτική εμπειρογνωμοσύνη και έρευνα ανάπτυξη και την στρατιωτική από την άλλη πλευρά, το στρατιωτικό σκέλος. Τέλος, υπάρχει και μια ρήτρα ραντεβού, που προτείναμε δηλαδή στους ηγέτες να επανέλθουν σε αυτό το θέμα και η ιδέα είναι να επανέλθουν το Δεκέμβριο του 2015 γνωρίζοντα ότι το καλοκαίρι του 2014 υπάρχει η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ οπότε δίνεται μια κάποια συνέχεια και ζητήθηκε να, να, να, να γίνουν προτάσεις. Τι έγινε, μακρηγόρησα, έχω ακόμα δύο λεφτά. Ναι. Ε, λοιπόν, πολύ σύντομα για τις αποστολές. Καταρχήν το Μαλί. Για να σας είστε νόμεροι, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αποστολή στο Μαλή κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει να κάνει πολλά ακόμα και χτες βασικά η PSC συμφωνήθηκε να παραταθεί για δύο χρόνια. Οι πολιτικές αποστολές που βρισκόμαστε τώρα εκεί, στο οποίο το συζητήσαμε χτες, υπήρξε κάποιο έγγραφο ενημερωτικό με ερωτήσεις προς τη ΣΥΦΚΟΜ με στόχο να επανέλθει στην PSC πριν το τέλος του έτους ώστε να ανατεθεί στις υπηρεσίες να αναπτύξουν ε, ένα σύευση, είμαστε σε ένα περαιτέρω στάδιο δηλαδή. Και εκεί στο Μαλί βέβαια μπήκε και ο ΙΕ που είναι κάτι το καλό, αλλά έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά την άφηξη του απαραίτητου προσωπικού. Νομίζω έχουν 9.000, 9.000 έπρεπε να είναι αφρικανικές δυνάμεις εκεί τα αφρικανικά στρατεύματα και είναι μόνο 4.000 για την ώρα. Υπάρχει πρόβλημα στην αστυνόμευση, αλλά αυτό είναι εκτελεστικό ζήτημα. Δηλαδή είναι έξω στου δρόμου, εμεί που, αυτό που θέλουμε να κάνουμε να εκπαιδεύσουμε και να φτιάξουμε το Υπουργείο Ασφαλείας για τη Σομαλία και εκεί η Αταλάντα ε, έχει κλείσει, αλλά η αίσθηση είναι ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε την επαγρύπνηση εκεί και παρετάθη για άλλα δύο χρόνια. Νέστορ, ε, δύσκολο να το ξεκίνημα. Τώρα νομίζω έχει κάπως μπει σε, μια, σε ένα δρόμο. Έχουμε νέο επικεφαλή τη αποστολή. Είναι πολύ σημαντικό ότι η έμφαση δίνεται περισσότερο τώρα στην επικράτεια της Σομαλίας. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι ίδιοι οι Σομαλοί να αναπτύξουν αστυνομικέ δυνάμεις. Ε, περισσότερο δηλαδή δίνουμε έμφαση στην ίδια τη Σομαλία και η UTM Σομαλία η κατάρτιση των σομαλικών ε, δυνάμεων ασφαλείας έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούμε πια να φτιάξουμε αυτόν τον σομαλικό στρατό. Γι' αυτό ναι. βέβαια πρέπει να είμαστε στο Μογκαντήσιο. Τώρα μετακινηθήκαμε και το περισσότερο προσωπικό είναι ήδη εκεί, ειδικά αυτοί που εργάζονται για τις δομές. Λιβύη, η πολιτική αποστολή στα σύνορα ε, υπάρχει κόσμος εκεί από το Μάιο. Ε, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ιδιαίτερα ε, παρόλα αυτά και παρά τις δυσκολίες δουλεύουν, αλλά βεβαίως είδατε ποια είναι η ασφάλεια εκεί. Τη μια, τη μια στιγμή απαγάγουν τον Πρωθυπουργό, μπούκαραν στο κτίριο το, όπου ήταν το ξενοδοχείο και πρώτη πόρτα δεξιά ήταν η δική μας αποστολή. Λίγο αργότερα έγινε ε, μια διαδήλωση. Κάποιοι από αυτούς τους ε, πολιτοφύλακες ε, αρχίσαν να πυροβολούν στο ψαχνό, 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολα, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικά, γιατί η σημαντική αυτή η αποστολή, γιατί συνδέεται με το θέμα της μετανάστευσης και της παράνομης μετανάστευσης. Ο κόσμος που έρχεται Οπότε η Βόρεια Αφρική δεν προέρχεται αναγκαστικά από τη Λιβύη. Πολλές φορές ε, έρχεται από την ή και ακόμη πιο μακριά. Είναι χώρα διέλευσης, οπότε ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε στα σύνορα αυτά θα είναι σημαντικό. Και υπάρχει και η πρόταση των Ιταλών να γίνει κάτι με την ΚΠΑ, μια αποστολή με τρεις επιλογές, μια στην ανοιχτή θάλασσα, μια να βοηθήσουμε τις χώρες στα σύνορα και τρίτον αυτή η οικοδόμηση δυνατοτήτων στις χώρες διέλευσης. Μια επιχείρηση στην ανοιχτή θάλασσα θα ήταν δύσκολο κάπως ε, από ό,τι κατάλαβα για τα κράτη-μέλη, αλλά ίσως ε, στην, ε, στην οικοδόμηση δυνατοτήτων να μην ήταν αδύνατη τέτοια συνεργασία. Για το ΚΑΡ, για την ΚΑΡ και την Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, ξέρετε και ακούτε ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση πια εκεί. Οι αφρικανικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν διευκόλυνση, τίποτα. Και μεταξύ έχουν όλο ένα και μεγαλύτερες ομάδες ε, ε, επαναστατών, ληστών, με όπλα που κάνουν ό,τι θέλουν. Οι Γάλλοι ενισχύουν την παρουσία τους εκεί, αλλά γίνεται και μια κίνηση εντός της Ένωσης, μήπως μπορούσαμε να στηρίξουμε. Και αυτό θα συζητηθεί αύριο στην PC. Ε, συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως, αλλά νομίζω πως ήταν σημαντικά όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομερείς αυτές τις πληροφορίες, τις χρειαζόμαστε. Αντιστράτηγε Φόσελ Σούμπερ. Παρακαλώ. Oh, came own. Uh, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να σας μιλήσω σε αυτό το διακεκριμένο ακροατήριο και θέλω να στηρίξω και εγώ αυτά που είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μου σχετικά με τις εκθέσεις και τις απόψεις που προέρχονται από τη δική σας την Επιτροπή κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τώρα μου προσφέρεται ευκαιρία να κάνω μια αναδρομή προς τα πίσω στους πρώτους έξι μήνες της ε, θητείας μου, να βγάλω τα πρώτα μου συμπεράσματα για το μέλλον και κατόπιν να βρω και μια ε, διασύνδεση με το πρώτο Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας που θα λάβει η χώρα το Δεκέμβρη. Ε, σε αυτούς τους έξι μήνες αυξήθηκαν κατά πολύ οι επιχειρήσεις λόγω των εξελίξεων που, υπήρχαν, που υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας. Συνεχίστηκαν λοιπόν οι αποστολές και επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση. Εγώ απλά θέλω να συμπληρώσω αυτά τα οποία ανέφερε ακροτηγός ο Βόλτερ για την Αταλάντα, για την επιχείρηση αυτή. Ε, συζητιέται να παραταθεί η αποστολή και επίσης ε, συζητιέται να χρησιμοποιηθούν στο βαθμό του δυνατού οι πόροι που έχουμε για να στηρίξουμε και τις άλλες αποστολές που έχουμε αναπτύξει στην περιοχή. Ε, την επιχείρηση Νέστορ ε, που αφορά στη Σομαλία και άλλες. Πρέπει να μείνουμε για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία. Αυτός είναι ο βασικός μας ρόλος και εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι η Σομαλία, το να περάσουμε στο Μογκαντήσο. Εδώ έχουμε δύο καθήκοντα. Το ένα είναι εξειδικευμένη εκπαίδευση και το δεύτερο είναι συμβουλευτικός ρόλος. Αυτά απέναντι στις ε, στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της ε, Σομαλίας. Βεβαίως θα είναι περισσότερο απαραίτητο να συντονιστούμε και με άλλους παίκτες, ε, κυρίως με άλλες αποστολές στην περιοχή. Όσον αφορά το Μαλί, γίνεται συζήτηση και εκεί για παράταση της αποστολής, διότι εξακολουθεί να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα που πρέπει να επιτύχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Μαλή έτσι ώστε η επιτυχία που σημειώσαμε στην εκπαίδευση να παραμείνει. Και αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται δύο πράγματα. Να εκπαιδευτούν περισσότερα στρατεύματα και δεύτερον να υπάρχει συνέχεια για εκείνες ε, τις μονάδες ε, που έχουν εκπαιδευτεί τώρα. Έχουμε δύο μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στο Μαλί και η τρίτη μονάδα πρόκειται να ολοκληρώσει σύντομα την εκπαίδευσή της. Ε, αυτά όσον αφορά τις αποστολές και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα διδάγματα που έχουμε βγάλει, θα αναφέρω ένα και μόνο. Ανακαλύψαμε ότι όσον αφορά τις ε, μη εκτελεστικές ε, εντολές, εκεί δεν έχουμε λειτουργική έδρα, άρα αυτοί αναφέρονται στα κεντρικά. Ας πούμε για την Αθήνα, για αυτό το πρόγραμμα. Είναι υπεύθυνη για την τέταρτη γενιά και για άλλα στρατηγικής φύσεως ε, θέματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Η UMS ε, στηρίζει όλα αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλα περισσότερα σχετικά. Επίσης, έχουμε όλο και μεγαλύτερο φόρτο στις συμβουλές που παρέχουμε, στο συμβουλευτικό μας έργο. Και αυτό φαίνεται κυρίως στις εξελίξεις που προέκυψαν στην ε, Αίγυπτο, στη Συρία, ε, στις μεταναστευτικές ροές και ας μην ξεχνάμε και τον κόλπο της Γουινέας. Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω, κυρίως σε σχέση με νέες διαδικασίες διαχείρισης ε, κρίσεων είναι ότι η, στρατιωτική τεχνογνωσία πρέπει να περιλαμβάνεται από την αρχή και σε όλη τη φάση του σχεδιασμού. Αυτό απαιτεί βέβαια να συγκεντρώνονται έγκαιρα οι πληροφορίες. Αναφέρομαι και σε πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ενημερώνουμε έγκαιρα το σχεδιασμό μας και να βασίζουμε την ανάλυση μας σε αυτό που μπορούν να πράξουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, επιθυμούμε να αφομοιώνουμε την στρατιωτική διάσταση καλύτερα σε αυτό το μηχανισμό τον ολοκληρωμένο μηχανισμό της υπηρεσία εξωτερικής δράσης που αφορά στις δικές μας αποστολές. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας. Εμείς, η δική μας επιτροπή, ε, θέλω να σας πω τι ακριβώς ε, πιστεύουμε σχετικά με τους ε, τρεις βασικούς τομείς που περιγράφηκαν πρόσφατα. Ο επικεφαλής της άμυνας έκανε παρατηρήσεις που είναι και οι προσδοκίες που έχουμε απέναντι στο Συμβούλιο και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν. Πρώτον, ε, το στρατηγικό περιεχόμενο που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρεται στο εισαγωγικό κομμάτι της έκθεσης. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε θέματα στρατηγικής. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά τα επόμενα έτη χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, με ποια ποιότητα και ποια ένταση. Επίσης, όλα αυτά πρέπει να εξαστούν κάτω από ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Οφείλουμε να εμβαθύνουμε και να βελτιώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια ανάμεσα σε όσους κάνουν το σχεδιασμό και μεγαλύτερη διαφάνεια επίσης ε, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Αναφερθήκατε στην ταχεία αντίδραση και είμαι ευγνώμων που αναφέρεται κυρίως ε, για τη συμμετοχή των ομάδων κρούσης. Ε, πράγματι ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στοιχεία τα οποία θα καθιστούν τις ομάδες κρούσης πιο ευέλικτες, πιο ευπροσάρμοστες καταστάσεις. Επίσης, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των κρατών μελών στην εκπαίδευση, ε, να υπάρχουν μεγαλύτερες περίοδοι εκπαίδευσης, να υπάρχουν καλύτερα εναρμονισμένα συστήματα για τις ομάδες κρούσης και για τα στοιχεία ταχείας αντίδρασης. Επίσης επιθυμούμε να προβάλλουμε περισσότερο τη στρατιωτική διάσταση σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της ε, θαλάσσιας ασφάλειας. Μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των θαλασσών, ε, η συνειδητοποίηση των καταστάσεων. Αυτά όλα έχουν στρατιωτική διάσταση και στις αρχές του επόμενου έτους όλα αυτά θα τα εξετάσουμε. Όσον αφορά τις συνεργασίες, η συνεργασία συνεχίζεται με το ΝΑΤΟ, εμβαθύνεται με τα Ηνωμένα Έθνη και με την Αφρικανική Ένωση. Αναφέρθηκε το Μαλί, είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης ε, για να μπορούμε να επιτυγχάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό. Και επίσης πάμε τώρα στον κρίκο με τον τρίτο τομέα. Ο επικεφαλής της άμυνας ανέφερε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εξελίξουμε περαιτέρω το, την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση. Χρειαζόμαστε ικανότητες από τα κράτη-μέλη και για να τις επιτύχουμε αυτές χρειαζόμαστε project. Project τα οποία τα ε, συντάσσει, τα φτιάχνει η βιομηχανία ή τα στηρίζει η βιομηχανία αν θέλετε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες εναντί του Συμβουλίου και θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσδοκία είναι να υπάρξει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σε θέματα άμυνας, να προβληθεί η στρατιωτική διάσταση στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και ολοκληρώνοντας θέλω να πω και ότι η συνέχεια είναι καθοριστική σημασίας. Το κενό από το Δεκέμβρη μέχρι το επόμενο Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου θα πρέπει κάπως να γεβηρωθεί με συναντήσεις benchmarking και συγκρίσεων που θα επιτρέψουν να διατηρηθεί ο ε, δυναμισμός και θα επιτρέψουν να μπορούμε να δούμε ε, σε κάποιο βαθμό κατά πόσον επιτύχαμε τους στόχους μας σε σχέση με το Συμβούλιο. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Ε, μας είπατε πολλές φορές ότι δεν πρέπει να έχουμε πολλές προσδοκίες από τη διάσκεψη κορυφής, αλλά έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Κοπά, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Σε σχέση λοιπόν με τις 70 ε, σελίδες που αναφέρατε, ε, πιστεύω πως τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι αναμέναμε. Ξέρετε ότι το επίπεδο προσδοκιών φιλοδοξιών του Κοινοβουλίου ήταν πολύ υψηλό. με τον κίνδυνο να είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά αυτό που θέλαμε ήταν να στείλουμε το μήνυμα πως η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει για μας η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου δεν θα πρέπει να είναι ένα γεγονός έκτακτο, θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια, θα πρέπει να είναι η αρχή και όχι το τέλος αυτής της συζήτησης που μέχρι στιγμή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα θέλαμε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης και κάποια ορόσημα και να γίνεται μια τέτοια συνεδρίαση όχι σε βάση ad hoc αλλά ας πούμε κάθε δύο χρόνια. Εάν πιστεύουμε, και νομίζω πως αυτό είναι κοινή άποψη, αν πιστεύουμε στα θέματα αμήνης, θα πρέπει αυτό να γίνει αισθητό και στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτό με οδηγεί στη δεύτερη μου παρατήρηση που αφορά την ορατότητα της ΚΠΑ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει μια ε, στρατηγική επικοινωνιακή απέναντι στο Συμβούλιο και τους άλλους ε, εταίρους. Γιατί Φυσικά είναι μια διαδικασία περιπλοκή που μένει σε επίπεδο ηγετών, αλλά εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες μας, γιατί είναι σημαντικό το θέμα, ιδιαίτερα σοβούσης της ε, τόσο σοβαρής οικονομικής κρίσης, ε, θα φανούμε άσχετοι και το θέμα το ίδιο. Και όπως ξέρετε είμαστε έξι μήνες πριν μια πολύ δύσκολη ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση όπου ε, κινδυνεύουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ε, είναι πολύ ακραίο και το αισθανόμαστε εδώ. Για όσους λοιπόν πιστεύουμε ότι το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι ένας από τους βασικούς τομείς ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, τότε θα πρέπει η επικοινωνία μας ε, με τους πολίτες να είναι καλύτερη. Ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κανεί σε κοινό παρονομαστή. Νομίζω λοιπόν πω εδώ τα πράγματα είναι σχετικά θετικά. Περιμένουμε και να δούμε τα επόμενα βήματα και σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σα εδώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Κοπά, ο κύριο Νταφ. Σα ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλου και ευχαριστώ του ομιλητέ μα για αυτά που εγώ πιστεύω ήταν ενθαρρυντικά. Αλλά θα πρέπει να πω πως εξακολουθώ να παραμένω προβληματισμένος όσον αφορά την δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεδομένου ότι έχει όλα αυτά τα άλλα πράγματα στην δέντα του, ορισμένα είναι πολύ κρίσιμα. Αμφιβάλλω κατά πόσο οι Πρωθυπουργοί μας θα αφιερώσουν αρκετό χρόνο και προσοχή σε αυτά τα πολύ σημαντικά και σοβαρά θέματα που τα συζητάμε εμείς εδώ όλο το απόγευμα και πρέπει κανείς να δει ότι οι Υπουργοί δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν για τα συμπεράσματα και τελικά υπεγράφησαν μόνο από το Συμβούλιο Νεότητος και Αθλητισμού τελικά από τους Υπουργούς δηλαδή Νεότητας και, και Αθλητισμού ε, για Επίσης πιστεύω πως είναι ένα μέγα σφάλμα τα απορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην αναφέρονται καθόλου στη συνεισφορά του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας, ότι τουλάχιστον από ευγένεια θα έπρεπε να αναφέρουν τη δικιά μας δουλειά, αλλά επίσης επειδή η δουλειά μας σε αυτό το θέμα ήταν εξαιρετικά καλή. Και νομίζω πως ε, θετικά και δημιουργικά διατυπώσαμε κάποια πράγματα και εκθέσαμε τους προγραμματισμούς για διάφορα θέματα και διάφορες επίμαχες καταστάσεις που οι ίδιοι οι υπουργοί δυσκολεύονται να το κάνουν. Οπότε παρακαλώ προσπαθήστε να μιλήσετε με το γραφείο του Φανρομπόη και θυμήσατε του την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να αυξήσει και την ε, αυξανόμενη ορατότητα ε, αυτού του θέματος για τον τύπο. Επίσης, βρίσκω σε αυτήν την ε, μακρά ε, παρουσίαση που έχουμε από πλευρά σας ότι δεν αναφέρεται παρακώς η αδυναμία των σχέσεων μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ. Για μας αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και κρίσιμο ότι δεν υπάρχει ροή δηλαδή ε, στις σχέσεις αυτές ε, δεν είναι αρκετά ε, ομαλές ώστε να έχουμε μια σοβαρή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα πρέπει η σχέση αυτή να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Περίμενα επίσης να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάγκη εξέβρεσης οικονομιών κλίμακας στους εξοπλισμούς καθώς και σχέσεις κόστος ωφέλειας περισσότερο από ό,τι έχουμε σε αυτό το έγγραφο και θα ήθελα να δω την έκφραση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο μεγαλύτερη έμφαση στο EDA που υπάρχει αλλά δεν αξιοποιείται αρκετά. Θα έπρεπε να αναβαθμιστεί. Και τώρα σε σχέση με τα ε, clusters, ε, τις ομάδες, ε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι λέει, εκείνοι θα πρέπει να δουν, εμείς θα πρέπει να δούμε. Πάντως να εξεταστεί η κατάλληλη χρήση των σχετικών άρθρων της συνθήκης. Ναι, πάρα πολύ ωραία, αλλά η συνθήκη ισχύει εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν έχουμε δει να προκύπτουν συγκεκριμένα σοβαρά κλάστερς ή ομάδες με αποστολές. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη. Πιστεύω πως το Κοινοβούλιο, Πρόεδρε, θα έπρεπε σοβαρά να σκεφτεί πώς εμείς θα ακολουθήσουμε και θα παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, δεν νομίζω πως ο κύριος Βαν Ρομπόη και η δική του παρουσίαση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα είναι κάποια επαρκής βάση για ποιοτική ανταλλαγή απόψεων. Ίσως λοιπόν να πρέπει να εφεύρουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ, Άντριου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να θυμίσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πως υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Άκουσα μάλιστα από κάποιοι λένε ε, ε ότι μας βλέπουν οι με μας τη νύχτα και ξυπνάνε στα μέσα της νύχτας και ουρλιάζοντας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τις ανησυχίες των Προελισάντων ότι οι πρωθυπουργοί τελικά δεν θα έχουν αρκετό χρόνο να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και επίσης ε, και ότι είναι δύσκολο να ε, συμμετάσχουν ε, ε, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη σε αυτά τα θέματα και όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί πριν από τη συνάντηση κορυφής. Θέλω όμως να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Στίβεν σχετικά με την Κεντρική Αφρική, τη δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Νομίζω η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πολύ, τα προβλήματα είναι οξύτατα και ρωτώ. Έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε εκεί τις ομάδες κρούσης και εάν ναι, Γιατί, ποια είναι τα επιχείρηματα υπέρ και κατά. Ο κύριος Τάνοκ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με την κυρία Κοπά ότι στην επόμενη θητεία το επόμενο κοινοβούλιο μπορεί να μην είναι τόσο φιλικά διακείμενο απέναντι σε αυτά προγράμματα όσο το τρέχον. Στη δική μου τη χώρα, κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πείσει τους πολίτε για την υπεραξία γενικά τη κοινή αυτή πολιτική. Ε, δύσκολο βέβαια αυτό και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίε ε, για επικαλύψει ε, και για το ε, κατά πόσον τον ε, αποκοπεί ε, κανείς από τον ΝΑΤΟ, κατά πόσον αυτό πραγματικά έχει μία αξία. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί είναι τρομοκρατημένοι με τον ιδέα του Ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα λάθος και γι' αυτό πρέπει να πείσουμε κυρίως Βρετανούς επί του θέματος. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Η έκθεση για το κέρες Αφρικής έγινε πέρυσι και εγώ ήμουνα μπλεγμένο σε αυτή αυτό το επιχείρημα υπέρ ή όχι της επιχείρησης Αταλάντα. Ο πρόεδρος της ήρθε στην Επιτροπή και ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, μείωση της ε, πειρατείας στην ακτογραμμή του. Τότε υπήρχαν υπόνοιε ότι κάποια από τα κονδύλια, τα χρήματα ε, της πειρατείας δόθηκαν στον Σαμπάμπ. Βεβαίως βελτιώθηκε το μεταξύ κατάσταση και διαρωτώ με γιατί η μείωση της πειρατείας συνδέεται συνδέεται με, την, με τον με την Κένια. Μήπως ε, θα πρέπει επίσης ε, να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως είπε και η κυρία Κρόμπερ και με κάπληψε για την Κεντρική Αφρική πριν από κάποιες ημέρες ήμουνα με την κυρία Τζόρτζοβα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ήταν πάρα πολύ ανήσυχη. Μίλησε μάλιστα και είπε ότι ε, θα μπορούσε να γίνει ένα, μια γενοκτονία τύπου Ρουάντας. Ε, εγώ δεν είδα βέβαια αυτή τη θρησκευτική διάσταση ανάμεσα στους μουσουλμάνους ε, και τους χριστιανούς, τα θύματα τους χριστιανούς, αλλά ερωτώ ποιες είναι οι δυνατότητες ε, στρατιωτικής επέμβασης. Θα μπορούσε να κινητοποιηθεί μία μάχημη ομάδα. Αυτά που έκαναν οι Γάλλοι στο Μαλί για να επέμβουν και να σταθεροποιήσουν τη χώρα. Τι είδους σκέψει υπάρχουν, γιατί άλλη μια Ρουάντα πιστεύω ότι θα ήταν ολέτριο και θα ήταν και μια μεγάλη αναστάτωση στην διεθνή κοινή γνώμη ότι δεν κάναμε τίποτα για να εμποδίσουμε την κατάσταση. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, ορισμένα σχόλια και κάποιες ερωτήσεις που απευθύνονται γενικά στους κυρίους, δεν είναι σε κάποιον συγκεκριμένο. Ε, καταρχήν η ομάδα μας και εγώ προσωπικά είμαι σφόδρα αντίθετος με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενδυνόμενη στρατιωτικοποίησή της. Και νομίζω υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα που μας επιβεβαιώνουν σε αυτή την αντίθεση. Παραδείγματο χάρη επειδή έγινε λόγο για το Μαλί. Ξέρετε γίνανε εκλογές ε, πρόσφατα. Πολύ χαμηλή συμμετοχή. Γιατί άραγε. Γίνεται λόγος τώρα για την κατάσταση που υπάρχει στην ε, Κεντρική Αφρική. Ποια είναι η αιτία της αστάθειας του προβλήματος. Λιβύη δεν, δεν μπορούμε να αφαιρεθούμε από το γεγονό ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι αποτέλεσμα ενό πολέμου στο οποίο συμμετείχε ενεργά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια εντυνόμενη αποσταθεροποίηση και μια ε, άσχημη κατάσταση για την οποία ευθύνεται και η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ζήτημα. Και από τα στοιχεία των ε, εκθέσεων που έχουμε δει και το έγγραφο της κυρίας Άστον και γενικά είναι προφανές ότι ανησυχούν πάρα πολύ οι αντιθέσεις και ανταγωνισμοί με Κίνα, χώρες BRICS, Ρωσία και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Είναι, είναι πασιφανές αυτό. Και αν θέλετε, όταν και εσείς μιλήσατε, αλλά όπως και ο κύριος Ντενζόν, στην τελευταία σύνοδο του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ζητήματα άμυνας, όπου επανέφερε μια θέση που με κάνει μεγάλη εντύπωση. Είπε ο κύριος Δενζόν ότι καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση μόνη της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της άμυνας. Και ρωτάω, για να γίνονται τέτοιοι ισχυρισμοί, δύο τι να συμβαίνουν. Είτε ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόσαστε, γιατί εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, να αντιμετωπίσετε μεγάλες δυνάμεις στις παγκόσμιες αγορές σε, έναν τέτοιο πόλεμο, οπότε καταλαβαίνω πραγματικά καμία χώρα μόνη της δεν σε θέση να, ή υπάρχει ένα άλλο θέμα, και αυτό έχει να ε, το λέω γιατί έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα battle groups. Καταλαβαίνουν οι κυβερνήσει των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουν όλο και λιγότερη διεθνή νομιμοποίηση για επιχειρήσει όπω είναι αυτή του Μάλι ή όπω είναι αυτή στη Σομαλία μόνε του και θέλουν μια συμμαχία με χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να φαίνεται ότι τη δράση αναλαμβάνει ένα διεθνή οργανισμό και όχι μια μεμονωμένη χώρα. Τώρα έρχομαι στο συγκεκριμένο ερώτημα για τα battle groups. Εμείς είμαστε αντίθετοι, σας το λέω, γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες οδηγούν στη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε έναν στρατιωτικό συνασπισμό, όπως είναι το ΝΑΤΟ και πιο επιθετικό ακόμα κατά τη γνώμη μου, γιατί εδώ θέλετε να υπάρχει και πολεμική βιομηχανία για αυτόν τον συνασπισμό, που δεν υπάρχει ενιαία στο ΝΑΤΟ. Αλλά, battle groups. Ποιο είναι ο λόγο που δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Εγώ έχω μια εξήγηση. Δεν χρησιμοποιηθήκαν γιατί διαφωνούν χωρισμένοι μεταξύ τους. Και διαφωνούν γιατί είναι, ε, δεν συμπίπτουν τα συμφέροντα. Είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και σου λέει γιατί να πάμε σε μια περιοχή που εμεί δεν έχουμε συμφέρον, α να δούμε. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα. Δεν μιλήσατε καθόλου για το pooling and sharing. Και ξέρετε, γενικά υπάρχει ένα θέμα. Ανοίγουν θέματα από το Συμβούλιο, από τον οργανισμό, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, από την Υπηρεσία Εξωτερική δράση δεν συζητούνται στον κόσμο, δεν εξηγούνται καν στο Ευρωκοινοβούλιο, ανοίγουν, κλείνουν, εξαφανίζονται. Pooling and sharing. Ωραία, έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Ρωτάω, το pooling and sharing δεν προϋποθέτει και αλλαγή των αμυντικών δογμάτων των χωρών μελών. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, παραδείγματο χάρη, να συμμετέχουν κάποιοι σε κοινού εξοπλισμού οι οποίοι όμω μετά δεν μπορούν να του χρησιμοποιήσουν, γιατί κάποιοι άλλοι προφανώ δεν θα συμφωνήσουν. Αυτό δεν προϋποθέτει να υπάρχουν κοινή αμυντικά δόγματα των χωρών μελών. Γύρω από αυτό το ζήτημα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Και τέλος, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας, πολεμική βιομηχανία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Ε, στο πρόβλημα της ε, πολεμικής βιομηχανίας, επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα, για μας είναι σαφές ένα ζήτημα. Όπως και οι άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το τομέα, κερδισμένες θα βγουν οι μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες. Χαμένες θα βγουν οι πολεμικές βιομηχανίες των μικρών χωρών. Και σας δίνω ένα παράδειγμα της Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κλείνει, κλείνουν όποιες μονάδες πολεμικής βιομηχανίας ε, υπάρχουν. Όλα αυτά βεβαίως στο όνομα της κρίσης, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Όμως υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που ε, αυτό αν θέλετε ξεπερνάει και μια κατάσταση που υπάρχει. Αν δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ε, ισότιμη συμμετοχή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη. Thank you very much, gentlemen. Ευχαριστώ πολύ κύριοι. Ε, πέντε λεπτά ο καθένας. Θέλετε εσείς ε, στρατηγία να αρχίσετε. Θα αρχίσω με το θέμα της στρατηγικής επικοινωνίας. Πράγματι, αυτό είναι κομμάτι των προσδοκιών μας. Θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για την στρατηγική επικοινωνία, όχι μόνο για το Συμβούλιο, αλλά και για τον ευρύτερο τομέα της CSDP. Κατόπιν, η ερώτηση για το Κοινοβούλιο αφορούσε εσένα. Τώρα, όσον αφορά τις, τα battle groups γενικά. Αυτή ήταν ε, ε, εν μέρη η διάγνωση για το, για το λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκαν προσπαθούμε να κάνουμε πιθανές βελτιώσεις για να γίνει πιο ευέλικτη η χρήση τους. Πάντως τελικά θα εξαρτάται από την πολιτική θέληση των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν ή να μην χρησιμοποιήσουν τα battle group και να συνεισφέρουν σε αυτά και να χρησιμοποιήσουν τα χωριστά τους στοιχεία, σαφώς. Όμως μπορούμε να διευκολύνουμε την πορεία αυτή με τυποποίηση, με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, όλες, όλα αυτά τα πράγματα ε, περιλαμβάνονται και στα συμπεράσματα και στα έγγραφα. Θα στραφώ τώρα στον όρο που χρησιμοποιήθηκε «Ευρωπαϊκός στρατός». Τίποτα στα έγγραφα δεν αναφέρεται κατά διάνοια σε ευρωπαϊκό στρατό. Ζητείται περισσότερη συνεργασία, αυξημένη διαφάνεια και όσο είναι δυνατόν αλλά και πάλι ανάλογα με την, ε, θα εξαρτηθεί αυτό από την επιθυμία των κρατών μελών περισσότερη κοινή δουλειά όσον αφορά την αντίληψη. Το ίδιο ισχύει για το pooling and sharing. Το pooling and sharing είναι ένα εργαλείο. Αυτό καθε αυτό δεν αποτελεί φιλοσοφία. Ήταν ένα εργαλείο ώστε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να χρησιμοποιούν τους οικονομικούς και υλικούς τους πόρους πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορεί να επιτευχθεί αυτό με άλλους τρόπους και ήδη έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα συνεργασίας για την εξοικονόμηση κόστους. Το pooling and sharing είναι επίσης ένα ευέλικτο εργαλείο. Μπορεί να ξεκινήσουμε από επίπεδα όπου να υπάρχει μια γενική ετοιμότητα, διάθεση χρησιμοποίηση. Ας πούμε η εκπαίδευση, οι ασκήσεις από εδώ και πέρα μπορούν να γίνονται μαζί χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, από τη δική μου πλευρά, τη στρατιωτική, επαναλαμβάνω και θέλω να πω ότι αυτό που χρειαζόμαστε από την εμπειρία μας από τις επιχειρήσεις, να υπάρχουν προϊόντα πάνω, με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, προϊόντα τα οποία να χρησιμοποιούμε διαλειτουργικά. Επανέρχομαι στην επιχείρηση στο Τσάντ, που από ό,τι θυμάμαι είχαμε όσα διαφορετικά μέλη συμμετείχαν, τόσα διαφορετικά ήταν και τα μαχητικά οχήματα. Εδώ λοιπόν οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρωθούν. Τώρα από τις στρατιωτική σκοπιά θα ήθελα να καταλήξουμε το εξή. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Έχουμε τακτικέ και πολύ συχνέ ε, ε, ανταλλαγέ και άτυπα και σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό που δεν έχουμε, αλλά αυτό αφορά το πολιτικό επίπεδο, δεν έχουμε τακτικέ, επίσημε επαφέ σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ αν θέλετε να μου επιτρέψετε να απαντήσω στι ερωτήσει του κυρίου Αγκουράκη. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Μαλί, να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικό τη Αφρικής, αλλά από ό,τι άκουσα η συμμετοχή δεν ήταν τόσο περιορισμένη, ήταν αρκετά καλή. Και πρέπει κανείς ε, να συγκρίνει βέβαια και με την κατάσταση που υπήρχε και τις εκλογές. Ναι. Νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, για συμμετοχή. Και για να είμαστε ειλικρινεί, αν υπάρχει ένα παράδειγμα όπου η διεθνή κοινότητα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν συμφωνήσει όλοι, ήταν αυτή. Ε, είχαμε τα Ηνωμένα Έθνη, ε, την Αφρικανική Ένωση, την ΕΚΟΑΣ, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπάθησαν να ορίσουν τι πρέπει να γίνει και να ακολουθήσουν όλοι και τη σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Γιατί ήταν ο στρατός που κανείς δεν τον υπολόγιζε, κάτι λοιπόν έπρεπε να γίνει. Κατόπιν τούτου, αν συγκρίνεται το τι υπήρχε πριν από ένα χρόνο και το τι υπάρχει σήμερα, ε, εντάξει δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Τώρα, κατά πόσον έχει στρατιωτικοποιηθεί η άμυνα ε, στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, τις δικές τους τις ε, στρατιωτικές δυνατότητες. Εμείς δεν τις αυξήνουμε. Λέμε βέβαια ότι ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση γιατί υπάρχουν όλο και μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα. Αν λοιπόν θέλουν να διατηρήσουν μια ικανότητα, τουλάχιστον την δική τους ικανότητα, γιατί υπάρχει αυτό, θα πρέπει να συνεργαστούν. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα πίσω από αυτά που ακούσαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν συμφωνίες με τη Ρωσία, με την Κίνα, μεγάλες συμφωνίες. Όχι, απλά κάθε κράτος να έχει αυτό που είναι σημαντικό και αυτονόητο να μπορεί να μείνεται και στη γειτονιά του. Γιατί βεβαίως μην ξεχνάτε, αν δεν μιλάς σε κανένα, δεν έχει κανείς τα μέσα και κανείς δεν σε υπολογίζει. Άρα δηλαδή αυτό επηρεάζει την κατάσταση ε, που επικρατεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο να συνεργάζονται οι δυνάμεις. Αλλά στη τελική ανάλυση, όταν φτάνουμε στη φάση ανάπτυξης των δυνάμεων, ξέρετε, το πιο αστείο είναι ότι έχει έχουν ήδη υπάρξει κάποιες ε, μάχημες ομάδες, τα battle groups που χρησιμοποιήθηκαν το 2003. Τότε στάλησαν τα battle groups για να προστατεύσουν μια πόλη ε, στην οποία είχαν επιτεθεί ε, αντάρτες, είχαν σκοτώσει ανθρώπους και μετά από αυτό υπήρχε η έννοια των battle groups και για να είμαστε ειλικρινείς όσοι βρίσκονται μέσα στα battle groups Βεβαίως υπάρχει και το ότι αν ας πούμε ε, μία, κάποιος από το βορρά είναι σε ένα battle group, ε, μπορεί να μην ενδιαφέρεται πολύ για την Αφρική. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και το θέμα του κόστους. Αν το στείλει κανείς για τρεις-τέσσερις μήνες πρέπει να καλύψει το κόστος. Άρα δηλαδή όσοι είναι μέσα στα battle groups δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την κάλυψη του κόστου. Άρα υπάρχει και το οικονομικό στοιχείο. Και αν υπήρχε μια καλύτερη ρύθμιση, αυτό θα ήταν σημαντικότερο. Αυτό όμω που είναι καθοριστικό είναι η πολιτική βούληση. Εγώ δεν μίλησα για pooling and sharing, δεν είπα αυτέ τι λέξει, αλλά αυτά που εννοούσα έχουν σχέση ε, με το pooling and sharing και πράγματι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην οτροπία και στο δόγμα, αλλά κυρίως στην οτροπία των ανθρώπων. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί όταν συγκεντρώνει και μοιράζεται κανείς πράγματα, υπάρχουν και χρονικά περιθώρια. Οι Βέλγοι, ας πούμε, πρέπει παραδείγματο χάρη να παραγγείλουν ένα αεροσκάφο. Η διάρκεια ζωή του είναι 10 χρόνια. Και όταν θα θελήσουν να συνεργαστούν με κάποιου άλλου, ε, να μην συμπίπτει η χρονική περίοδο. Ο χρονισμός λοιπόν είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσον αφορά τη βιομηχανία, είδαμε ότι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για το ότι οι μεγάλοι εποφελούνται περισσότερο από τους μικρούς και σε αυτό ασκήσαμε πίεση. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν καινοτομίες, να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να υπάρχουν και θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρώπης και μερικοί λένε ότι και εμείς θέλουμε ε, να συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Υπάρχουν παλιές βιομηχανίες που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές και που θέλουν να τις προστατεύσουν. Νομίζω όλα αυτά εμπλέκονται στη συζήτηση. Και αναφέρουμε στη συζήτηση που θα έχουν οι ηγέτες. Τώρα, κατά πόσον θα υπάρχει αρκετός χρόνος, βεβαίως ε, ενδέχεται να μην υπάρχει ε, πολύς χρόνος ε, γιατί υπάρχει το θέμα της ε, τραπεζικής ενοποίησης ε, και πολλά άλλα. Αλλά εν το έχουν υποσχεθεί. Καταρχήν, το σημαντικότερο είναι ότι θα μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, άρα δηλαδή νομίζω ότι έχουν πιστεί ότι θα πρέπει να έχουν κάποιο χρόνο για να συζητήσουν τα θέματα, τουλάχιστον δύο ώρες. Ο κύριος Μπαρομπέι είναι ε, πεπισμένος και όπως είπε και η κυρία Κοπά, οι, υπουργοί ξέρουν ότι δεν θα είναι μια και έξω, θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια και να αναφέρεται στα συμπεράσματα ε, το τι συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Το κοινοβούλιο ε, κατά πόσο ήταν φιλόδοξο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι φιλόδοξο το κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει να βλέπουν τι είναι ρεαλιστικά εφικτό. Τα συμπεράσματα ε, πρέπει να είναι φιλόδοξα αλλά και ρεαλιστικά. Ίσως έχετε δίκιο όσον αφορά ε, στους εταίρους κυρίως ε, στο ΝΑΤΟ ίσως εκεί η γλώσσα να έπρεπε να είναι διαφορετική αλλά πρέπει να έχετε κατά νου ότι όσον αφορά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην διάμεση έκθεση και την τελευταία έκθεση της κυρίας Άστον έχουν υπάρξει παρεμβάσεις από πολλούς και από τον ΝΑΤΟ που επιθυμούν να συνεργαστούν. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ίσως λοιπόν τώρα για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα και η Νότιος Κορέα να συμμετάσχει σε μία από τις αποστολές μας. Κατά πόσο είναι απαραίτητο, κοιτάξτε, δείχνει κάποιο ενδιαφέρον και μπορούν να συνδεθούν και αυτοί με το πρόγραμμα Νέστορας και με την πειρατεία. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον. Υπάρχουν ε, πολλοί εταίροι που ενδιαφέρονται ε, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι και τα άρθρα της συνθήκης ε, δεν είναι απόλυτα διαφανή. Νομίζω αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν συμφωνούν πάντα ε, για το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Για το Στάρντοκ υπάρχει η πολιτική βούληση και υπάρχουν πράγματα τα οποία ήδη υφίστανται ο μηχανισμός Αθηνά. Ίσως ε, και το θέμα της ε, χρηματοδότησης ε, των πολιτικών αποστολών. Και από αυτού πρέπει να υπάρχει σαφής διατύπωση. μπορούμε να δούμε και το τι, πώς ακριβώς θα διατυπώσουμε και το ότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη συνεχώς να συμβάλλουν. Δεν ακούω βέβαια να το θίγουν αυτό τα κράτη-μέλη. Νομίζω στην αρχή το συζήτησαν οι υπουργοί και αυτό που βλέπω να υπάρχει τώρα είναι περισσότερο περιφερειακά κλάστερ. Τα βλέπει κανείς αυτά και στο ΝΑΤΟ, αυτά τα μορφώματα. Όσον αφορά την Αταλάντα, την πειρατεία, την Al-Shabaab, Κοιτάξτε και πάλι δεν είμαι ειδικό, αλλά εγώ από ό,τι έχω καταλάβει υποτίθεται αυτόματα τα χρήματα από την πειρατεία πάνε στην Al-Shabaab. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, γιατί ε, δεν είναι τόσο δομημένη όλη αυτή η σχέση. Σίγουρα υπάρχουν πολλά δίκτυα πίσω από την πειρατεία και εάν δεν προσέξουμε ε, ενδέχεται να εξαπλωθεί. Ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά χρειαζόμαστε αποφάσεις δικαστηρίων για να μπορέσουμε να τους διώξουμε. Η al είναι άλλο πρόβλημα, γιατί αυτοί ελέγχουν μεγάλα κομμάτια της Ομαλίας. και το μόνο όπλο που έχουμε εναντίον είναι η Άμισον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για την Άμισον. Τώρα οι Κενιάτες γίνονται πιο δραστήριοι, του ζητήθηκε να αυξηθεί η συμμετοχή τους. Υπάρχει λοιπόν δυσκολία να βρούμε τα χρήματα. Επίσης, οι Άμισομ ε, έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν είναι σωστά εξοπλισμένοι, δεν έχουν ας πούμε ελικόπτερα, δεν μπορούν να μετακινηθούν τόσο γρήγορα. Βεβαίως, οι μεγαλύτεροι εγγύηση που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι που έχουμε εκπαιδεύσει εντάσσονται στην Άμισομ, όμως δεν έχουν συγκεκριμένη ε, δομή. Ε, αυτά είχα σε μεγάλο βαθμό να πω. Ε, και μία ερώτηση για την δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Τζορτζέβα ήταν στην πίση η Επίτροπος και πρέπει να σας πω ότι ανησυχήσαμε κι εμείς ε, πάρα πολύ. Ίσως θέλετε τι είπε ο ε, αναπληρωτής ε, γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που δεν μίλησε για γενοκτονία αλλά και αυτός χρησιμοποίησε πολλά σκληρά λόγια. Και επίσης από επιτόπου πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει έχουμε καταλήξει στο ότι η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. παλαιότερα δεν υπήρχε το θρησκευτικό στοιχείο, τώρα όμως έχει παρισφρήσει και αυτό. Επιδεινώνεται λοιπόν η κατάσταση. Οι Γάλλοι πρόκειται να στείλουν ε, περισσότερες ε, μάχημες ομάδες και εμείς ε, σκεπτόμαστε το αν θα πρέπει να στείλουμε battle groups. Αυτό ως δυνατότητα επιλογή συμπληρωματικά προς αυτά που κάνουν οι Γάλλοι. Υπάρχουν λοιπόν επαφές, αλλά αύριο θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και νομίζω πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ε, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή η συζήτηση θα γίνει αύριο. Και κατόπιν ε, θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε τις επαφές μας με τα Ηνωμένα Έθνη και με άλλους, με τους Γάλλους. Εκεί μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά αναφερθήκατε στην Πούνια, νομίζω ότι και εκεί μπορεί να υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Αυτό ακόμα δουλεύει μαγειρεύεται, να δούμε λιγάκι τι πιστεύουν τα κράτη-μέλη. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει πρόβλημα και όσο καθυστερούμε ε, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται το πρόβλημα. πολλοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα ξεφύγει ε, από έλεγχο και μετά θα κατηγορηθούν αυτοί που ασχολούνται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Υπάρχει και ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και η Αφρικανική ε, Ένωση δεν κάνει τίποτα, ίσως γιατί αυτοί δεν έχουν ε, καμία δυνατότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε στην Υποεπιτροπή Το Τελευταίο μου καθήκον είναι να σας θυμίσω ότι η επόμενη ε, συνάντησή μας θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Θα είναι και η τελευταία μας για φέτος. πέρα συνεδρίασης. Thank to